Καλημέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί μας περιορίζει ο χρόνος και έχουμε και ακρόαση σήμερα το πρωί. Ας μην καθυστερούμε περισσότερο. Να σας πω ότι αποφάσισαν οι συντονιστές χτες στη συνάντησή τους. Έχουν μοιραστεί. Θα τα έχετε δει. Οπότε αν έχετε αντιρρήσει να τι πείτε, Αλλιώ εφόσον δεν πείτε καμία αντίρρηση, εγκρίνονται οι αποφάσει αυτές. Και περνάμε στην ακρόαση. Όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατίας της Κορέας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ τους φιλοξενούμενους μας, τους προσκεκλημένους μας, που έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέμα και μεγάλη γνώση στο διεθνές εμπόριο. Ζητάω από τους ομιλητές να περιοριστούν στις αρχικές τους παρατηρήσεις σε 10 λεπτά. Γιατί έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να προχωρήσουμε και σε συζήτηση στη συνέχεια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω εγώ στην εισαγωγή μου, θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον κύριο Στίβεν Βόλκοκ. Εδώ. Ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο London School of Economics σε θέματα ε, διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Και εγώ ήμουνα τη δεκαετία του 70 μαθητής εκεί, φοιτητής. Μετά Μάλλον πρώτα θα δώσω τον καθηγητή Βούλκοκ το λόγο και μετά θα προχωρήσουμε στους επόμενους. Ευχαριστώ. Να σας στήσω και τον συνάδελφό μου, τον Ζαν ο ε, έχει συνεισφέρει στην μελέτη αυτή. Και πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια μελέτη η οποία έγινε από το συντονιστικό σώμα του ΕΛΕΣΥ, e, το ΣΕΠΣ e και το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ και το Deutsche Wirtschaft, το Γερμανικό Ινστιτούτο. Έχουμε βασιστεί σε ήδη υπάρχον υλικό, δεν έχουμε κάνει καινούργιες έρευνες, για να αξιολογήσουμε κάπως ισορροπημένα λοιπόν τη δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά την συμφωνία αυτή με την Κορέα. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κορέα λοιπόν προσφέρει μια ευκαιρία για ελεύθερες συναλλαγές πέρα από άλλες συμφωνίες όπως είναι η Core US, η συμφωνία δηλαδή, της Κορέας με τις ΗΠΑ που δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Είναι μια συνολική συμφωνία, ίσως η πιο πλήρης που έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα από πλευράς της Κορέας. Υπάρχει μεγάλη ελευθέρωση στα αγαθά, στις υπηρεσίες και η συμφωνία έχει και κάποια καινούρια στοιχεία όσον αφορά τις διατάξεις. Για το θέμα της συμβατότητας με τον ΠΟΕΜ, μας ζητήσατε να το κοιτάξουμε αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία νομίζω ότι υπάρχει πλήρη συνοχή. Δεχόμαστε δηλαδή τις ερμηνείες ε, του ΠΟΕ όσον αφορά τα άρθρα 24 του ΓΚΑΤ και 5 του ΓΚΑΤΣ για τα δασμολογικά εμπόδια και άλλες διατάξεις. Άρα λοιπόν η συμφωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΠΟΕ όσον αφορά το εμπόριο. Αυτό που κάνει η συμφωνία είναι ότι θέτει σε εφαρμογή τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του ΠΟΕ, και φροντίζει για ερμηνευτικές διατάξεις και εφαρμοστικές διατάξεις. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου η συμφωνία είναι ΠΟΕΣΥΝ σε τομείς όπως είναι ο ανταγωνισμός για παράδειγμα επειδή δεν υπάρχουν διατάξεις στον ΠΟΕ όπως επίσης για τις δημόσιες συμβάσεις και εκεί είναι μάλλον ΠΟΕ συν ή GPA συν. Ίσως κυρίως για τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπου ξεπερνά τη συμφωνία TRIPS σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τους γεωγραφικούς δείκτες, όπου βάζει δύο ε, μητρώα και ευθυγραμμίζεται με αυτά που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα αυτό. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχει βέβαια κάποια αμφισβήτηση για το πνεύμα της πολυμερούς συμφωνίας και γίνεται συζήτηση για το κατά πόσο η... το περιεχόμενο των πολυμερών συμφωνιών συνάδει όχι με τη συμφωνία αυτή. Πάντως, οι διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι το κύριο μέσο που χρησιμοποιείται για εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Όσον αφορά τα ωφέλη, πρέπει να σας πω ότι τα σχόλιά μου βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες μελέτες. Δεν έχουμε κάνει εμείς καινούριε μελέτες. Το φέλη λοιπόν είναι περιορισμένα κάτω από 1% του ΕΠ για την Κορέα και κάτω από το 0,1% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κορέα αποφελείται περισσότερο επειδή είναι μια πιο μικρή οικονομία και επειδή η Κορέα έχει υψηλά επίπεδα προστασίας μέχρι τώρα. Τα στοιχεία αυτά για μας είναι καλά. Πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε το Μάιο που μας ε, πέρασε. Οπότε νομίζω ότι είναι σωστά τα ποσά που αναφέρουμε εδώ. Οι εμπορικές επιπτώσεις τώρα. Όλο και περισσότεροι τομείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν από τις εξαγωγές παραχάνουν. Υπάρχουν μεγάλα ωφέλη και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και όσον αφορά την μηχανική, τη φαρμακευτική, τη χημική βιομηχανία και σε έναν βαθμό και η γεωργία και τα τρόφιμα, γιατί έχουν περισσότερες εξαγωγές. Η πιο πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως λέει ότι έχουμε 33 δις κέρδος στις εξαγωγές ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι είναι η σωστή τάξη μεγέθους αυτή, γιατί είναι παραπάνω από ό,τι μας λένε προηγούμενες μελέτες, αλλά αυτή η πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μπει περισσότερο σε λεπτομέρειες και προσπαθεί να εκφράσει ποσοτικά τα κέρδη από το εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη και τους δεσμολογικούς φραγμούς που υπάρχουν. Βέβαια, το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δεν θα άρει τα μη δασμολογικά εμπόδια, μπορεί να καταργήσει τους δασμούς, αλλά όχι τα μη δασμολογικά εμπόδια. Εδώ θέλει παραπάνω δουλειά. Άρα τα ωφέλη αυτά εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό από τα αποτελεσματικά μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των μη δασμολογικών φραγμών. Εμπορικές επιπτώσεις για την Κορέα και πάλι χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία όσον αφορά τα κέρδη της Κορέας από τις εξαγωγές είναι 23 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει λιγότερο από το έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κορέα. Βέβαια η μελέτη δείχνει ότι περιορίζονται τα κέρδη στην αυτοκινητοβιομηχανία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σε ένα βαθμό και στην υφαντουργία και την ηλεκτρονική. Στην υφαντουργία πολύ λιγότερο βέβαια όσον αφορά τον όγκο των εξαγωγών. Όλες οι μελέτες πάντως και οι πιο πρόσφατοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις ξένες επενδύσεις της Κορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Τσεχία και την Σλοβακία, για παράδειγμα. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις όσον αφορά το επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αλλαγή και στον όγκο των εξαγωγών της Κορέας. Πάντως τώρα τα duty drawback, οι διατάξεις δηλαδή σχετικές ε, με τις επιστροφές δασμών, το duty drawback, αν κοιτάξουμε τις διάφορες εκτιμήσεις που υπάρχουν ε, για τις συνέπειες, έχουμε 1,5% του κόστους αν αυτοκίνητο. Αν δούμε τώρα το θέμα των ε, ρυθμίσεων, των κανόνων για τους μη δεσμολογικούς ε, φραγμούς. Οι διατάξεις είναι πολύ σημαντικές εφόσον κερδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας μάλιστα και ρυθμίσεις ανατομέα για την αυτοκινητοβιομηχανία, για τις μηχανές, τη μηχανική και φάρμακα. Αυτοί οι διακανονισμοί που γίνονται λοιπόν ανακλάδο, ανατομέα, προσφέρουν καλές προοπτικές και αντιμετωπίζουν τις ε, μέχρι τώρα διατάξεις για τα TPD που υπήρχαν μέχρι τώρα στην Κορέα. Και οι Κορεάτες χρησιμοποιούν κάτι αντίστοιχο. Έχουν μια νέα έννοια του moderator third party. Και έτσι εξετάζουν τις περιπτώσεις όπου έχει μια διαφωνία υπάρχει κάτι σαν διαιτησία. διατάξεων, διακανονισμού, επίλυσης διαφορών. Όπως προβλέπεται και στη Συμφωνία Κόριους, δηλαδή Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, όπως είπα και πριν, είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τον συνολικό στόχο για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Συμπεριλαμβάνει τα δύο μητρώα που έχουμε, τους γεωγραφικούς δείκτες και είναι TRIPS SYN. Αν λάβουμε υπόψη μας ε, τις διατάξεις που αναφέρονται σε παραβάσεις σε κλιματικού χαρακτήρα. Και σε άλλους τομείς ξεπερνάει τη συμφωνία TRIPS για τον ανταγωνισμό. Υπάρχει μια παράλληλη συμφωνία διμερής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κορέα για συνεργασία και εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα περιλαμβάνει και διατάξεις για τη διαφάνεια που ανήκει στον ΠΟΕΣΥΝ. Για τις δημόσιες συμβάσεις τώρα, ακριβώς επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα έχουν υπογράψει συμφωνίες ε, για αγορές, Εδώ έχουμε προσθέσει κάποιες υποχρεώσεις στον τομέα των αγορών από την Κορέα για τέτοιες συμβάσεις. Οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με την επίλυση διαφορών περιλαμβάνουν διαφορές τύπου παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου με μια διαδικασία γρήγορη. Για την εφόρο ανάπτυξη τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε το περιβάλλον και με τις συνθήκες εργασίας, οι συμφωνίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν διατάξεις που ε, προωθούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές εργασίας και η Κορέα αναλαμβάνει τη δέσμευση για αξιοπρεπή εργασία. Υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές που έχουν να κάνουν ε, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και που δεν έχει επικυρώσει ακόμα η Κορέα. Αλλά η συμφωνία λέει ότι δεσμεύονται τα δύο μέρη να συμμορφωθούν με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες συμβάσει του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Υπάρχουν και εδώ πάντως διαδικαστικά μέτρα που προβλέπονται και που θα διευκολύνουν την πρόθεση προδιαγραφών για την εργασία βάσει του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Για το θέμα τώρα του χρονοδιαγράμματος. Εδώ υπάρχει το θέμα κατά πόσο αν θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά γρήγορα η συμφωνία. Λέμε στην εκθεσή μας ότι υπάρχουν κάποια πλονεκτήματα ήδη από την αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες αλλά και την ε, μηχανική υπέρ. Δηλαδή θα αποφεληθούμε από αυτά εφόσον γρήγορα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία και όχι αν καθυστερήσει. Τελικά θα έλεγα ότι η συμφωνία αυτή είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες έχουν τα υπέρ και τα κατά, έχουν και κάποιο κόστος, αλλιώς δεν θα πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, αν υπολογίσουμε το κόστος που χρειάζεται για την προσαρμογή από μια τέτοια συμφωνία, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ λίγο, αν συγκρίνουμε μάλιστα με άλλες συμφωνίες. Χρειάζονται κάποιες προσαρμογές σε ορισμένους τομείς ή υποτομείς που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία αυτή. Πάντως, αν κατακλείδη να σας πω ότι η αύξηση των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέψεων NTB. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ο δεύτερος μας ομιλητής είναι ο Ιγνάσιο Γκαρθία, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, μόνιμος καλεσμένος στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην συνεδρίασή μας, κύριε Ιγνάσιο Γκαρθία. Παρακαλώ μην ξεπεράσετε τα δεκάλεπτα κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ο Ντέβιτ Σάλιβαν λυπάται ειλικρινά που για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παραστεί στη δημόσια αυτή ακρόαση όπως θα ήθελε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το ΕΛΕΣΥ e για την ποιότητα αυτής της μελέτης που εκπώνησε, που είναι πολύ περιεκτική και μεστή. Εγώ θα περιοριστώ σε τέσσερα μόνο σημεία στην δική μου ομιλία και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά το δυναμικό σε ό,τι αφορά το first mover advantage του πλεονεκτήματος για την πρώτη αυτή κίνηση, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες και στη μεταπητική βιομηχανία. Οι τέσσερις βασικές μεταπητικές βιομηχανίες είναι τα μηχανήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκινητοβιομηχανία και χημικά προϊόντα. Στους τέσσερις αυτούς τομείς οι δασμοί που εφαρμόζει η Νότια Κορέα είναι αρκετά υψηλή, μεταξύ 6 και 8%. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, υπάρχει πολύ σημαντικός ανταγωνισμός με άλλε χώρε του ΩΣΑ, ιδιαίτερα την Ιαπωνία και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Σε όλους αυτούς τους τέσσερις τομείς που σας προανέφερα, οι δασμοί για τις ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές ε, θα καταργηθούν ε, σταδιακά μέσα σε μία τριετία. Οπότε υπάρχει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, πλεονέκτημα, first mover advantage, εξαιτίας της σταδιακής κατάργησης των δασμών που προβλέπει η συμφωνία αυτή ελευθερία Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι το θέμα των μη δεσμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, και στην φαρμακοβιομηχανία ή στην παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων, όλες, όλοι οι μη δεσμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο που έχουν εντοπιστεί από τους αρμόδιους κλάδους είναι τομείς που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τη συμφωνία το θέμα των μη δεσμολογικών φραγμών. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο βασικό μη δεσμολογικό φραγμός είναι ότι η Κορέα εφαρμόζει μια, ένα πολύ περίεργο συνδυασμό αμερικανικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Για να ε, τεθεί σε εμπορία ένα προϊόν στην αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί στι συγκεκριμένε και αυστηρέ προδιαγραφέ που εφαρμόζει η Κορέα, κάτι που αυξάνουν το κόστος ε, και επιβαρύνουν πολύ τον παραγωγό και πάρα πολλέ προδιαγραφέ, περιβαλλοντικέ και ασφάλεια δημιούργησαν ένα είδο μη δεσμολογικών φραγμών. Τώρα πια η Κορέα αναγνώρισε την ισοδυναμία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών με τι κορεατικέ. Οπότε μειώθηκε αυτό ο μη δεσμολογικό φραγμός. Για τα ηλεκτρονικά προϊόντα, ο μη δεσμολογικό φραγμό οφείλεται στο πολύ επιβαρημένο ρυθμιστικό καθεστώ που εφαρμόζει η Κορέα, που υποχρεώνει ε, την ε, εξέταση και πιστοποίηση από ένα τρίτο μέρος. Αυτό ευτυχώς καταργήθηκε και τώρα ελαφρύθηκε ο ρυθμιστικός ε, μηχανισμός που εφαρμόζει η Κορέα και είναι παρόμοιος πια με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τους μελλοντικού δεσμολογικούς φρεγμούς υπάρχουν κάποιε νομικά δεσμευτικέ διατάξει για την αποτροπή αυτών των κινδύνων και προβλέπει και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό διακανονισμού των διαφορών. Ιδιαίτερα στην το βιομηχανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα σε 75 μέρες θα έχουμε μια α, ανεξάρτητη απόφαση τρίτου μέρους που θα αποφαίνεται για το κατά πόσο η Κορέα έχει σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Έτσι επιταχύνονται οι διαδικασίες και είναι πολύ πιο βραχές οι προθεσμίες από ό,τι στη Συμφωνία της Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι αφορά ε, και τα ηλεκτρονικά και τα προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας. Πολλές ε, δικές μας διατάξεις στη συμφωνία με την Κορέα δεν ε, Περιλαμβάνοντα την αντίστοιχη συμφωνία τους με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά συνάψαμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με ασιατική χώρα και η χώρα αυτή έχει δεχτεί την ρυθμιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει για τα αυτοκίνητα, για τα ηλεκτρονικά προϊόντα, για τους γεωγραφικούς δείκτες, αλλά και για πολλές άλλες πτυχές αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Τρίτον, η συμφωνία αυτή νομίζω ότι συνιστά με ένα πολύ σωστό τρόπο αντιμετώπιση και των εργασιακών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ακροθυγό τα ανέφερε και ο Στίβεν Γουλκοκ. Εγώ θα επιμείνω σε ένα σημείο κύριο και θα το διευκρινίσω. Σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, σε σχέση με τις συμβάσεις ε, της ε, ΔΟΕ, έχουμε τρία επίπεδα δεσμεύσεων. Καταρχήν, μια προσπάθεια ε, κύρωσης των συμβάσεων της ΔΟΕ, δέσμευση αποτελεσματικής εφαρμογής των ε, συμβάσεων που έχουν κυρωθεί και σε περίπτωση που δεν έχουν κυρωθεί κάποιες συμβάσεις της, ΔΟΕ, θέλουμε τουλάχιστον οι συνθήκες ε, οι εργασιακές να τηρούν την, τις συμβάσεις της ΔΟΕ του 1979. Αυτές είναι δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κορέα σε σχέση με τι προδιαγραφέ τη Διεθνού Οργάνωσης εργασία. Και μάλιστα η παρακολούθηση τη συμμόρφωση αυτών των διατάξεων θα αναμίξει άμεσα και την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή οι συνδικάτα, εργοδότε και μη κυβερνητικέ οργανώσει για πρώτη φορά θα εκπροσωπούνται άμεσα στον έλεγχο αυτή τη συμμόρφωση. Θα ήθελα επίση να πω δύο λόγια διάφορα, για διάφορα ευαίσθητα σημεία. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχαμε επίγνωση των ευαισθησιών της ευρωπαϊκής πλευράς και προσπαθήσαμε όλες αυτές οι ευαισθησίες ε, να ληφθούν υπόψη και να καλυφθούν από τη συμφωνία. Θα επιμείνω και εδώ σε τρία σημεία. Καταρχήν, μεταβατική περίοδο για την κατάργηση των δεσμών στις πιο ευαίσθητους τομείς. Είναι αρκετά ε, μακρά η περίοδος, είναι πενταετία. Επίσης, δεν υπήρξε σημαντική ελάφρυση των ε, ευρωπαϊκών κανόνων για την προέλευση. Σε ό,τι αφορά την ρήτρα διασφάλισης, προσπαθήσαμε να τη συμπεριλάβουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε περίπτωση που ανακύψουν. Φυσικά με τη διαδικασία συναπόφασης που προβλέπεται θα γίνει μια αξιολόγηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι θα βρούμε αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα ανακύψουν. Αυτά Νομίζω ότι η μελέτη του LSE και του καθηγητού Γουλκόκ έδειξε ότι το θέμα του duty drawback, της επιστροφής των δασμών, είναι ένα θέμα που από οικονομική άποψη δεν είναι τόσο σημαντικό αν το συγκρίνουμε με τα τεράστια ωφέλη που θα αποκομίσουμε από τη σύναψη της συμφωνίας με την Κορέα. Ευχαριστώ. Thank you, Ignacio. Ευχαριστούμε, Ιγνάσιο. Δεν χρησιμοποίησες ε, και τα 10 λεπτά. Τρίτος μας ομιλητής, ο κύριος Ιβαν Χόντακ, Γενικός Γραμματέας ε, του Συνδέσμου Ευρωπαίων Αυτο... Ε, Κατασκευαστών Αυτοκινήτων με σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες και στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Μπρούζ. Έχετε το λόγο κύριε Χόντακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που μου δίνεται την ευκαιρία για ακόμη μία φορά να παρουσιάσω τη δική μας θέση για το σχέδιο της συμφωνίας με την Κορέα. Καταρχήν να πω πολύ σύντομα ότι το γεγονός ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμη η συμφωνία δείχνει ότι όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα και ξέρουμε ότι τα βασικά προγράμματα είναι, βρίσκονται στον ε, τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οπότε δεν σας λέω κάτι καινούριο. Επίσης, εκτιμούμε πάρα πολύ τη μελέτη που έγινε από το London School of Economics και θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσοχή σας στο ότι εδώ μιλούμε για ένα μείγμα ε, του υλικού που ήδη υπάρχει, μια δηλαδή συλλογή των στοιχείων που ήδη υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια νέα αξιολόγηση επιπτώσεων. Καταρχήν, να σας ε, δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για τη βιομηχανία. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 36,6% όλων των εργαθέσεων εργασία τη Ευρώπη έρχονται από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είτε συνδέονται άμεσα είτε έμεσα με τον τομέα αυτό. Έχουμε δηλαδή 10 εκατομμύρια εργαζόμενους στον τομέα αυτό και αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη με την παρούσα κατάσταση και τις ε, μεγάλες, ε, τα, οι μεγάλες τάσεις στην αυτοκινητομηχανία, όπως ξέρετε όλοι, ε, μας έχουν κάνει να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιο ανταγωνισμό, Κίνα, ασιατικές χώρες, Βραζιλία, ε, Ιαπωνία, όλες αυτές οι χώρες δεν είναι απλώς ανταγωνιστές, αλλά προστατεύουν και τη δική τους αυτοκινητοβιομηχανία. Το βλέπουμε και θα το δούμε να γίνεται και στο μέλλον. Ήδη με, τις, με, την, με Ινδία υπάρχει μια τέτοια ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ε, και με την Κίνα θα υπάρξει επίσης. Όλοι προσπαθούν να προστατεύσουν τον τομέα τους, τον κλάδο τους. Αλλά βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό, ε, σημαντική αυτοκινητοβιομηχανία και μεγάλο μερίδιο για την οικονομία. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μέσω και των διαπραγματεύσεων που γίνονται για τις ε, συμφωνίες αυτές η βάση των, ε, της κατασκευής ε, μεταφέρεται εκτός Ευρώπης και αυτό δημιουργεί προβλήματα για την βιομηχανία και για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, για τις υποχρεώσεις της κτλ. Τώρα πάμε στην συμφωνία για, με την Νότια Κορέα. Όλοι ξέρουμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας το... και ο τομέα αυτός είναι ένα τομέα βασικό για τι διαπραγματεύσει. και θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει μια καλή συμφωνία για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι κορεάτε ποτέ δεν θα υπέγραφαν την συμφωνία αυτή. Ένα είναι αυτό. Αυτό το έχει καταγράψει και ο κορεατικό τύπο και η βιομηχανία και οι αρχέ τη Όλοι το γνωρίζουν. Έχουμε δασμούς που θα, αφομοιωθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Κορέα και βεβαίως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνάψουμε τη συμφωνία με την Κορέα, αλλά θέλουμε να έχουμε μια ισόρροπη συμφωνία. Και πιστεύουμε ότι αυτή, η στιγμή, αυτή τη στιγμή η συμφωνία αυτή δεν είναι ισόρροπη. Ναι, η Κομισιόν έχει δίκιο, τα, οι μη δεσμολογικοί φραγμοί έχουν απαλληφθεί και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό, αλλά Υπάρχει μια πιθανότητα οι κορεάτε να εισαγάγουν νέου, δασμούς, νέου φραγμούς και αν δείτε τι ρήτρε διασφάλιση που υπάρχουν δεν μα δίνουν καμία εγγύηση ότι οι κορεατικέ αρχέ, ότι η κυβέρνηση τη Κορέα, δεν θα θέσει νέου φραγμού στο εμπόριο. Και ήδη το βλέπουμε αυτό και στι διαπραγματεύσει. σήμερα για την ε, νέα δομοθεσία που θα αφορά και τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ο τομέα λοιπόν αυτό είναι πραγματικά τομέα κλειδί για τι διαπραγματεύσει και ήταν και το διαπραγματευτικό χαρτί για, το, για τη δική μας βιομηχανία. Τώρα, αν δούμε την αγορά των καταναλωτών. Ανοίγουμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων για την Κορέα. Και αυτοί ανοίγουν για μας μια αγορά 49 εκατομμυρίων ατόμων. Η αυτοκινητοβιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 49 εκατομμύρια, 1,34 στην Κορέα, παραγωγή 40 εκατομμύρια στην Ευρώπη, 3,7 στην Κορέα εξαγωγές συνολικές οχημάτων 3,4 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 εκατομμύρια από την Κορέα. Οι διμερείς λοιπόν εξαγωγές αυτοκινήτων και ο μέσος όρος τα τελευταία 4 χρόνια είναι 32.500 αυτοκίνητα που πάνε από την Ευρώπη στην ε, Κορέα 541.500 που πάνε από την ε, Κορέα, που έρχονται από την Κορέα εδώ. Οι εξαγωγέ από Ευρώπη προ Κορέα είναι το 1% των συνολικών εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα αυτοκίνητα. Είναι 25% όμω για του κορεάτε το ποσοστό αυτό. Οπότε βλέπετε πόσο σημαντικό είναι ο τομέα αυτό. Οι ασυνέπειε και ανισορροπίε είναι σαφεί και στο, έλλειμμα, στο, στο έλλειμμα εμπορικού συζυγίου με την Κορέα. Μιλούμε για 14 δισεκατομμύρια. Η Eurostat μα τα έχει δώσει αυτά, 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι το 25% του συνολικού έλλειμματος. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν και τη δική μας αξιολόγηση, αυτό το έλλειμμα θα, μεγαλώσει, θα αυξηθεί ε, αναλογικά και με, τις, ε, με τα αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν στην αξιολόγηση της Κομισιόν. Νομίζω δηλαδή περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στον τομέα αυτό, ανοίγουμε τον τομέα και δεν κάνουμε τίποτα για να υπάρξει μια ισορροπία στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Το πρόβλημα λοιπόν θα μεγαλώσει. Αθέμητος ανταγωνισμός. Όπως είπα, η βιομηχανία αυτή δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ελεύθερες συναλλαγές και υποστηρίζουμε και την, ε, τον κύριο της Ντόχα, υποστηρίζουμε το άνοιγμα της αγοράς κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τον ανταγωνισμό. Πιστεύουμε ότι λόγω ακριβώς ε, του duty drawback που έχει δοθεί στους Κορεάτες και που δεν έχει δοθεί ποτέ σε κανένα άλλη χώρα του ΩΣΑ, δημιουργεί τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Οπότε ζητούμε το duty drawback να σταματήσει μετά από την πάυση των δασμολογικών των δασμών μετά τους, την απαλυφή των δασμών για να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των σχέσεών μας θα πρέπει να καταργηθεί το duty drawback από τους Κορεάτες. Γιατί ούτως ή άλλως η Ευρώπη δεν το έχει δώσει σε κανένα, σε καμιά άλλη χώρα του όσα. Και πέρα από αυτό θα, θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο για μελλοντικέ ε, συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών που θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα αριθμητικά στοιχεία τώρα για το duty drawback και τι σημαίνει είναι ε, διαφορετικά. Αλλά βασιζόμενοι στις ανεξάρτητες μελέτες που έχουν γίνει από την Credit Suisse, και αν ε, έχετε υπόψη σας και μια μεσαία ας πούμε, τιμή ενός αυτοκινήτου για 10.000 ε, ευρώ που εξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το duty drawback θα μπορεί να φτάσει 300 με 500 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο. Η Κομισιόν πρόσφατα είπε σε, ένα, σε μια συνέντευξη στην Frankfurter Allgemeine ότι ο στόχος ε, της, ε, της συμφωνίας αυτής με την Κορέα δεν ήταν να ανοίξει η ε, αγορά της ε, Κορέας για μικρά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Αλλά αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει, γιατί, αφού το κάνουμε αυτό, γιατί δεν γίνεται και το αντίστοιχο για εμάς. Και το άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι οι ρήτρες διασφάλισης. Διμερής ρήτρα διασφάλισης, η οποία θα πρέπει να μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα να σταματήσουμε τις ε, εισαγωγές, να λάβουμε άμεσα μέτρα. Δεν θεωρούμε ότι η ρήτρα διασφάλισης έτσι όπως είναι είναι λειτουργική και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι είναι πολύ περιορισμένη χρονικά. Και δεν χρειάζεται να είναι περιορισμένη χρονικά. Γιατί δηλαδή περιορίζουμε στα 10 χρόνια. Η ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και η ρήτρα διασφάλισης σίγουρα δεν ισοσκελίζει την, ε, τις ε, συνέπειες που υπάρχουν με σχέση με το duty drawback που έχει η Κορέα. Οπότε θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη σε μελλοντικέ συζητήσεις ε, που ελπίζουμε να υπάρξουν να ξεκαθαρίσουν τον ορισμό του τι δημιουργεί κάποιο πλήγμα, να, να δούμε τι γίνεται και με τις έρευνες. Βέβαια έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες η Κομισιόν ήδη να δώσουμε όμως και το δικαίωμα στην βιομηχανία να ζητήσει την εκπόνηση μιας έρευνας και από ό,τι κατάλαβα θα γίνει αυτό και υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Οπότε πρέπει να δούμε ε, προσεκτικά τη διμερή ρήτρα διασφάλισης. Επίσης, το ειδικό, την ειδική ρήτρα για το duty drawback που υπάρχει, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η ρήτρα να είναι λειτουργική γιατί προς το παρόν δεν είναι. Αν δούμε την αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν και κλείνω σε ένα λεπτό πρόεδρε, η Κομισιόν λέει, η αξιολόγηση μάλλον επιπτώσεων λέει ότι η βιομηχανία δεν θα κερδίσει από, την, από αυτή τη συμφωνία ελεύθερου συναλλαγών με την Κορέα, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις ή οι ασυνέπειες ε, θα αυξηθούν για ακόμα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι λέει η αξιολόγηση επιπτώσεων και η απασχολησιμότητα στην ε, ε, Ευρώπη θα πέσει κατά 1,5%. 1,5% στον τομέα της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας όμως μιλά, σημαίνει 30.000 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει κλείσιμο 10 εργοστασίων. Αν θέλετε να μεταφέρετε την κατασκευή έξω από την Ευρώπη, ένας τρόπος είναι αυτός. Αν θέλετε να κρατήσετε την ε, κατασκευή εντός της Ευρώπης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι ισόρροπη και όχι να είναι ισόρροπη μόνο για τις υπόλοιπες βιομηχανίες αλλά και για την ευρωπαϊκή αυτοκινητόβιομηχανία. Η ε, αξιολόγηση επιπτώσεων λέει ότι θα υπάρξει αύξηση 400% εξαγωγών από την Ευρώπη στην Κορέα μέσω της συμφωνίας. Αυτό δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει ποτέ. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθο εκεί που έγραφε 400 στο κείμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τρόπο ή καμιά πιθανότητα να υπάρχει τέτοια μεγάλη αύξηση 400 μονάδων προς, εξαγωγών προ την Κορέα. Και τέλο, ε, μη δεσμολογική φραγμή Πρέπει να έχουμε μία πολύ ισχυρή πιθανότητα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Κορεάτες δεν θα θέσουν νέους δασμούς, νέους τέτοιους φραγμούς και, και πρέπει να το εξασφαλίσουμε από την ε, συμφωνία αυτό. Γιατί προς τον παρόν η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στους Κορεάτες να, να βάλουν νέους φραγμούς μη δασμολογικούς και για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Ε, ελπίζω να υπάρξει όντως μια πιο ισόρροπη ε, συμφωνία. Καλώς. Ήσασταν ιδιαίτερα διεξοδικός. Το λόγο έχει τώρα ο Δόκτωρ Πασκάλ Καρνέης, ε, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Υπηρεσιών. Είναι ειδικευμένο ε, στο κοινοτικό δίκαιο. Έχει εργαστεί ω ε, νομικό σύμβουλο και εμπειρογνώμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ευρωπαϊκής Ενωσπονδίας Τραπεζών από το 1999 και είναι διαχειριστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρήσεων. Έχετε το λόγο κύριε Κερνέης. Ένα δεκάλεπτο παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Εν είδη παρουσίαση, ήθελα να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υπηρεσιών είναι, ένας οργανισμός, είναι μια οργάνωση που εκπροσωπεί σχεδόν όλους τους κλάδους των υπηρεσιών. Και Μιλούμε για, την ασφάλεια, για τις ασφάλειες, για να σας... Θα ήθελα παρακαλώ να σταματήσουν οι δυτικέ συνομιλίε στη διάρκεια των παρουσιάσεων. Τουλάχιστον οι δυτικέ συνομιλίε να γίνονται σιγανά και όχι χειρά γιατί εμποδίζουν τον ομιλητή. Συνεχίστε κυρία Κενέση. Ασφάλεια, τραπεζικές υπηρεσίε. Ε, διαμεσολάβηση σε ασφάλειες, διάφορα γεωργικά επαγγέλματα, μεταπητικές, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, κατασκευαστικός κλάδος, ε, ταχυδρομικές, υπηρεσίες delivery, ε, υπηρεσίες συναφής με το περιβάλλον, με την ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές, έχουν κέρια και νευραλική σημασία για την οικονομία. Ξέρουμε ότι οι υπηρεσίες ε, είναι θεμελιώδης για την οικονομία. Μιλήσαμε για την αυτοκινητοβιομηχανία που είναι σημαντική, αλλά μην ξεχνάτε ότι και στις υπηρεσίες 60% του συνολικού ΑΕΠ προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα στις υπηρεσίες. Ο ιδιωτικό τομέας ε, αντιπροσωπεύει 60% των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και 65% της απασχόλησης στην Ευρώπη αφορά απασχόληση στο ιδιωτικό φορέα στις υπηρεσίες. Πάνω από 100 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Δύο στου 10 εργαζόμενου στην Ευρώπη εργάζονται σε μια διεθνή δραστηριότητα υπηρεσιών. Οπότε οι υπηρεσίε για το διεθνέ εμπόριο είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Η νέα συμφωνία εμπορίου με την Κορέα είναι σημαντική και για τι υπηρεσίε και είναι γλαφυρά τα στοιχεία. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι εξαγωγέ αυξήθηκαν πάνω από 42%. Η Κορέα ήδη είναι πολύ σημαντικό εταίρο μα στι υπηρεσίε. Είναι ο ένατο εμπορικό μα εταίρο και η τάση μάλιστα θα συνεχίσει την αναδική τη πορεία τα επόμενα χρόνια. Αν ρίξουμε μια ματιά στο καθαρό πλεόνασμα της δικής, του δικού μας κλάδου με την Κορέα, βλέπουμε ότι αυξήθηκε από 2,3 δις το 2004 σε 2,5 3,5, ε, δηλαδή 1,2 δις επιπλέον ε, κέρδος ε, μέσα σε λίγα χρόνια. Πάνω από 50% δηλαδή αύξηση. Προσβλέπουμε σε μια συνέχιση, επαναλαμβάνω, αυτή τη ανωδική ε, τάση. Και ελπίζω ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα ενισχύσει αυτή την αναδική τάση και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουμε από το εμπόριο στις υπηρεσίες με την Κορέα. Ε, υπολογίζουμε με βάση τα 50% τη τελευταία πενταετίας, 10% το χρόνο περίπου αύξηση. Για να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η συμφωνία για το εμπόριο και μόνο για το καθαρό πλεόνασμα. Ήδη επαναλαμβάνω η τάση ανωδική είναι 10% το χρόνο. Η Eurostat είπε σε μία από τις μελέτες της ότι το εμπόριο με την Κορέα είναι χαμηλότερο. Η τάση για την Κορέα είναι χαμηλότερη από την τάση με τον υπόλοιπο κόσμο που είναι 12%. Πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ε, εναγωνίως αυτή τη συμφωνία για να αυξήσουμε αυτή την αυξητική τάση και στην περίπτωση της Κορέας και να καταλήξουμε σε μια αύξηση του καθαρού πλεονάσματος με την Κορέα της τάξης 15%, δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρό πλεόνασμα με την Κορέα. Αυτό θα είναι υποφελές φυσικά για το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώ. Και θα μας δώσει ένα καθαρό κέρδος μετά από μια πενταετή εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτη αυτή η εξέλιξη, γιατί ε, όσο περνάει η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μια ανάκαμψη και να καλύψουμε το χαμένο έδαφο στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τι υπηρεσίε όπω και για του άλλου τομεί και ευελπιστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κορέα. Οι υπηρεσίε ε, δεν αφορούν μόνο το διασυνοριακό εμπόριο. Οι υπηρεσίες αφορούν και τις ε, άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις. Προτιμούμε να πηγαίνουμε επί τόπου και να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στον τόπο τους, στην πατρίδα τους. Οπότε ε, δημιουργούμε κάποιες συμπράξεις ε, ή θηγατρικές στις χώρες. Αυτά για τις άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Κορέας μία επίσης ανωδική σημαντική τάση και μάλιστα την τελευταία πενταετία η Ευρώπη έχει επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ στη Νότια Κορέα. Βέβαια δεν είναι αρκετά γνωστό ότι οι επενδύσει αλλοδαπού εμπορίου, 74% του συνόλου των επενδύσεων που γίνονται προς την Κορέα γίνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτά είναι πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Μέχρι στιγμής η Κορέα δεν είχε καλή θέση από άποψη προσέλκυση ε, επενδυτικού κεφαλαίου από την Ευρώπη. Είναι ο ένατος εμπορικό εταίρος στι διεθνεί εμπορικέ εμπορικές συναλλαγές, αλλά είναι 16ος εταίρος μόνο για τι υπηρεσίε, Κάτι που δείχνει ότι εξακολουθούν να ορθώνονται πολλοί φραγμοί, ιδιαίτερα στι υπηρεσίε, που εμποδίζουν τι επιχειρήσει μα επιχειρήσεις μας να συνάψουν εμπορικέ συμφωνίε με την Κορέα. Οπότε η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου είναι πολύ σημαντική και από αυτή την άποψη, γιατί θα βελτιώσει... Ε, με εντυπωσιακό τρόπο τις δυνατότητες των επιχειρήσεών μας να έχουν συναλλαγές με την Κορέα. Οπότε η, ε, ο Ευρωπαϊκό Κλάδο των Υπηρεσιών είναι αναφαδόν υπέρ τη σύναψη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κορέα. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε το μήνυμα τη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και άλλων μεταπητικών κλάδων και αναλα... αντιλαμβανόμαστε τι ανησυχίε του. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ των ρητρών διασφάλιση και ελπίζω να το εξετάσει αυτό το Κοινοβούλιο ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού. Ζητούμε όμω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια σωστή αξιολόγηση του συνολικού πλεονεκτήματο αυτή τη συμφωνία, των συνολικών ωφελών. Να εξετάσουμε το τεράστιο δυναμικό και το τεράστιο πλεονέκτημα που θα δημιουργήσει η συμφωνία αυτή για τι ε, υπηρεσίε, για τον ευρωπαϊκό κλάδο των υπηρεσιών και άρα για το σύνολο τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που αναφέρθηκε από τον ε, καθηγητή του LSE είναι ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό προηγούμενο για παρόμοιε συμφωνίε ελευθέρω εμπορίου που θα συναυθούν στο μέλλον. Και μάλιστα δρομολογούνται, αλλά και στη γενική στρατηγική και στη μελλοντική μα εμπορική πολιτική, τέτοιε συμφωνίε και με άλλε χώρε. Αν δεν κυρωθεί η συμφωνία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω ε, κόλλησε στο Κογκρέσο στι ΗΠΑ η αντίστοιχη, τότε το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πληγεί, αλλά και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα δώσει μια κακή εντύπωση αξιοπιστίας. Έχουμε πάρα πολλές ε, συμφωνίες που δρομολογούνται, Σιγκαπούρη, Μεξικό, Μερκοσούρ κτλ. Γι' αυτό επίσης η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα μας δώσει και το πλεονέκτημα του first mover στην κορεατική αγορά. Της πρώτης σόδου, γιατί αν είμαστε οι πρώτοι που θα αποκτήσουμε τις άδειες, που θα καρποθούμε το μερίδιο του λέοντος στην καλύτερη θέση στην κορεατική αγορά, τότε θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα και τον ανταγωνισμό. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα ωφελήσει όχι μόνο τις υπηρεσίες, αλλά θα μας εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά και πλήρη εθνική μεταχείριση στην κορεατική αγορά. Θα εξασφαλίσει λοιπόν και τις επενδύσεις μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους επενδυτές και για τους ε, ηθήνοντες που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Οι διαπραγματευτές Κορέας ε, συμφώνησαν να δώσουν ε, ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αντίστοιχες με τις κορεατικών. Στις, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον μεταπητικό κλάδο, στα ηλεκτρονικά, στον τουρισμό και σε παρόμοιες κλάδους υπηρεσιών υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ ευρωπαϊκών και ερωτικών ε, επιχειρήσεων. Βέβαια, κάποιοι τομεί παραμένουν κλειστοί, αλλά η πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι στιγμή είναι εντυπωσιαστή. Γιατί σε ό,τι αφορά τα GATS, ε, σε σχέση με το γύρο του, της που είναι οι συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για μας, ε, ε, η Κορέα τότε είχε πολύ κακές επιδόσεις. Στο μεταξύ όμως, στην αναθεωρημένη προσφορά που έκανε στο GDA, στις διαπραγματεύσεις του ΓΚΑΤΣ, σημείωσε πρόοδο. Βέβαια έχουν αποτελματωθεί εκεί οι διαπραγματεύσεις, αλλά η αναθεωρημένη προσφορά ΓΚΑΤΣ της Κορέας είναι η βάση για τις νέες διαπραγματεύσεις. Και αν δούμε τι έδω πρόσφερε η Κορέα σε άλλους εμπορικούς εταίρους που ανταγωνίζονται τις δικές μας επιχειρήσεις, για παράδειγμα η Συμφωνία κόρου με τι Ηνωμένε διαπιστώνουμε ότι σχεδόν σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών που, που η συμφωνία που εξετάζεται σήμερα δίνει ένα κόρους συν σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες. Πολύ καλύτερες δηλαδή οι συνθήκες για μας από ό,τι για τους Αμερικανούς. Έτσι μπορούμε προοδευτικά να διεισδύσουμε σε τομείς υπηρεσιών που μέχρι στιγμής ήταν στεγανή και κλειστή στην κορεατική αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα οι δικηγόροι, για παράδειγμα, είναι τομέα που έχουν ε, τέτοιε νέε ανανεωμένες δυνατότητες. Βέβαια υπάρχει ένας φόβος ε, ε, να, να μην τηρήσει τις υποχρεώσει τη. Γι' αυτό και υπάρχει η δυνατότητα ρήτρε αναθεώρηση που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, γεφυρώνονται τα χάσματα και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα μπορούσα να αναφέρω ξεχωριστά τον κάθε τομέα, αλλά σας, έστειλα διεξοδική ανάλυση του κάθε τομέα των υπηρεσιών. Οπότε το μήνυμα είναι παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακυρώσει και να εφαρμόσει τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Νότια Κορέα το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. The next, ε, Ο επόμενος, αλλά πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, πρέπει να σας πω ότι οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες από τους ομιλητές μας και είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής αυτής. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ρενέ Φαν Σλότεν, που είναι Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας. Έχει μάστερ στην οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Κρόνιγκεν και από την Πρού, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο εκεί. Από το 1990 είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας. Κύριε Φανσλότεν, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Από ό,τι φαίνεται η δικιά μου η παρουσίαση δεν είναι παρουσίαση γιατί δεν βρίσκω εδώ τα slides, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που προσκάλεσε τη χημική βιομηχανία να έρθει εδώ στην ακρόαση αυτή όσον αφορά τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Όταν τον Οκτώβριο που μας πέρασε ξεκίνησε η συμφωνία αυτή, η χημική βιομηχανία εξέδωσε ένα ανακοινωθέν τύπου με το οποίο καλωσόριζε την συμφωνία αυτή και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ε, συμφωνία έτσι όπως έγιναν οι διαπραγματεύσεις και συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαίρετη αυτή συμφωνία που πέτυχε όσον αφορά τη χημική βιομηχανία. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας πόσο σημαντικό είναι το διεθνές εμπόριο για μια βιομηχανία όπως είναι η χημική. Είμαστε υδρογενής ε, βιομηχανία, παράγουμε χιλιάδες προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με ένα σωρό άλλα προϊόντα. Δεν μπορείτε να έχετε ανταγωνιστική φαντουργία, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικών. Όλα αυτά χρησιμοποιούν τη χημική βιομηχανία. Χημικά. Οπότε είμαστε η μητέρα της βιομηχανίας. Χωρίς εμάς δεν μπορείτε να έχετε μια σύγχρονη κοινωνία. Οπότε θέλω να σας δείξω, αν μου επιτρέπετε, πόσο σημαντικό είναι το εξωτερικό εμπόριο για τον κλάδο μας από το 1995 μέχρι το 2009 όσον αφορά τις εσωτερικές ε, συνολικές πωλήσει στην εσωτερική αγορά και στην εξωτερική. Θα δείτε ότι στο εσωτερικό από 58% έχουμε φτάσει στο 126% ενώ βλέπετε συγχρόνως πόσο σημαντική είναι εσωτερική αγορά για την χημική βιομηχανία. 27% το 95% και με τεράστια αύξηση το 2009. Βλέπετε επίσης τις πωλήσει τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες που από 15% το 95% έχουν φτάσει 26% το 2009. 25% των πωλήσεών μας πηγαίνουν σε εξωτερικές αγορές. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ελεύθερο εμπόριο, το ελεύθερο εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο μας, προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε άλλες αγορές. Οι εμπορικές ροές τώρα, ποιες είναι με τις κύριες εμπορικές ε, περιοχές. Ναύτα για παράδειγμα που αποτελεί στοιχείο κλειδί. Η Ασία επίσης είναι ένα σημαντικός προορισμός για τα προϊόντα μας. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν εδώ είναι ότι το εμπόριο με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι 50 δις ευρώ. Αλλά να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς βάζουμε δασμούς στο εμπόριο με τους πιο σημαντικούς εμπορικούς μας εταίρους. Οπότε, αν σκέφτεστε ότι από αυτά τα 50 δις έχουμε ένα 3% μέσο όρο δασμών, σημαίνει 1,5 δις σε δασμούς που πληρώνεται για το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι 1,5 είπαμε δισεκατομμύρια. Το 1 τρίτο τώρα όλων των χημικών εμπορικών συναλλαγών είναι εσωτερικό, σημαίνει ότι 500 εκατομμύρια πληρώνει ο κλάδος για να μπορεί να έχει εμπόριο στο εσωτερικό. Η Κορέα τώρα είναι μια πολύ σημαντική αγορά. Όσον αφορά τις πωλήσει είναι ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, σε βαθμό σημασίας. Βέβαια, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελεί μια αγορά κλειδί και η Κίνα, τη οποίες η σημασία αυξάνεται συνεχώ. Η Γερμανία, η Ιαπωνία επίση είναι σημαντική εταίρη. Είναι αυτέ που βρίσκονται στο top 30. Η Κορέα βρίσκεται και αυτή μεταξύ αυτών. Τώρα, το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κορέα, πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις εισαγωγές. Αγνοήστε λίγο το σημείο εκείνο που πέφτουν πάρα πολύ. Το 2009 οι εξαγωγές και οι εισαγωγές εξαιτία της κρίσης Πάντως έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εμπόριο με την Κορέα. Που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στην κορεατική αγορά. Τι εξάγουμε τώρα στην ε, Νότια Κορέα. Εξάγουμε κυρίως οργανικά χημικά πολυμερή, πετροχημικά, κυρίως πετροχημικά όμως και τα παραγωγά τους. Ας πούμε ότι αυτό είναι το τμήμα των πιο σημαντικών μας εξαγωγών προς τη Νότια Κορέα. Όσον αφορά τις εισαγωγές, θα δείτε ότι εισάγουμε από τη Νότια Κορέα κυρίως πολυμερή. Η Νότια Κορέα έχει έναν πολύ ανταγωνιστικό τομέα στα πολυμερή. Οπότε και εμείς περιμένουμε ότι εδώ θα έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό από την Κορέα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πάντως, θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς, η χημική βιομηχανία, δεν φοβόμαστε αυτόν τον ανταγωνισμό. Το ελεύθερο εμπόριο για μας είναι κάτι από το οποίο μπορεί να αποφεληθεί η βιομηχανία μας, ο κλάδος μας. Και σας εξήγησα γιατί. Αν ελευθερώσετε το εμπόριο στα χημικά, η πρώτη βιομηχανία που θα αποφεληθεί είναι ακριβώς η ίδια βιομηχανία. Διότι δεν παράγει κανείς όλα τα χημικά από μόνος του. Μειώνοντας λοιπόν το κόστος εισαγωγών, γιατί τότε πέφτει το κόστος των εισαγωγών με μια τέτοια συμφωνία, υποφελείστε κι εσείς και πιο πολύ μάλιστα. Όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι το ελεύθερο εμπόριο στη χημική βιομηχανία είναι κάτι θετικό. Η Κίνα για παράδειγμα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, διότι με την ένταξη στον ΠΟΕ προχώρησε σε τέτοιες συμφωνίες κάτι το οποίο έδωσε τεράστια όθηση στην χημική τους βιομηχανία, αλλά και όχι μόνο. Γιατί χρειάζεται τα χημικά η βιομηχανία γενικώ. Οπότε έτσι είναι ανταγωνιστική μια χώρα. Οπότε και μια χώρα που όπως είναι η Ινδία για παράδειγμα παραδοσιακά κλειστή, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να είναι αυτόνομη στα χημικά, θέλει και εκείνη ε, Τέτοιε συμφωνίες. Άρα λοιπόν οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλους. Η ελευθέρωση του εμπορίου στα χημικά λοιπόν πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται στα πλαίσια του ΠΟΕ. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ κολλάνε πολλές φορές, οπότε μέσα από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών βλέπουμε ε, μια δυνατότητα να πάμε ακόμα πιο πέρα από ό,τι πάμε στον ΠΟΕ. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτέ τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών κατά τη γνώμη μα. Εμεί δεν θέλουμε τέτοιε συμφωνίε με οποιαδήποτε χώρα. Η προτεραιότητα πρέπει να δίνουμε στι χώρε εκείνες που έχουν πραγματικά μεγάλο οικονομικό δυναμικό. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο των δασμών ή των μη δασμολογικών φραγμών. Πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη μα τι κίνδυνο υπάρχει εφόσον αποκλειστούμε από μια αγορά. Όταν κάποιο άλλο μεγάλο εταίρο έχει συνάψει τέτοιου είδου συμφωνία. Για παράδειγμα, τι έγινε μετά τη συμφωνία ναύτα όσον αφορά το εμπόριο με το Μεξικό. Ακριβώς επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν πρόσβαση ελεύθερη στην μεξικανική αγορά, χάσαμε το δικό μας μερίδιο στην αγορά αυτή. Άρα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται με τους εταίρους μας. Η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, η Κίνα, ε, η ΑΣΕΑΝ, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Ουκρανία, όλες αυτές είναι χώρε η Μερκοσούρ, που πρέπει να κοιτάμε. Δεν πρέπει όμω να φοβόμαστε τον ανταγωνισμό ούτε από τι ΗΠΑ ούτε από την Ιαπωνία ούτε πουθενά. Ο ανταγωνισμό έχει βοηθήσει την χημική βιομηχανία. Μα έχει εκθέσει στην παγκοσμιοποίηση πλήρω. Συγχρόνω όμω μα βοήθησε να γίνουμε περισσότερο καινοτόμοι, πιο αποτελεσματικοί και όσον αφορά τη χρήση ενέργεια. Οπότε πρέπει να δούμε ποιους εταίρους επιλέγουμε, να δούμε τι κάνουν οι άλλες χώρες, να ισχύουν οι κανόνες για την ε, χώρα καταγωγής. Είναι κάτι καλό πιστεύω στις συμφωνίες. Το παράδειγμα της Κορέας μας δείχνει ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σπάνε συμφωνίες ε, στο τέλος. Από την αρχή να είναι ξεκάθαρο δηλαδή τι σπάει τη συμφωνία και τι δεν τη σπάει. Από την αρχή να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και για την κατάργηση όλων ε, των μη δασμολογικών ε, φραγμών. Επίσης, να χρησιμοποιούνται οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών για να αντιμετωπίζουμε θέματα επιδοτήσεων, ε, διπλής τιμολόγησης, φορολόγησης εξαγωγών κλπ. Έτσι λοιπόν, είμαστε υπέρ της συμφωνίας αυτής. Θέλουμε να αρχίσει να ισχύει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι μια καλή συμφωνία. Καλύπτει πολλούς τομείς, όχι μόνο την πρόσβαση στις αγορές, αλλά και τις, επιδοτη... τι, συγγνώμη, και επενδύσεις και την ε, πνευματική ιδιοκτησία και άλλα. Όντω, ορισμένα σημεία στα πολυμερή, για παράδειγμα, όπω είπα και πριν, είμαστε πιο ευάλωτοι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίω διαπραγματευόμενη για τα πολυμερή, για την ελευθέρωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και μετά να αποδώσουμε καλύτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ελευθέρωση. Αυτή η συμφωνία αποτελεί και ένα καλό σήμα που στέλνουμε προς τους άλλους μας εταίρους. Για αλλιώ θα νομίζουν ότι δεν μπορούν να βασιστούν στην Ευρώπη οι εταίροι μας. Ευχαριστούμε. Τελευταίος μας ομιλητής, ο κύριος Ρόλαν Σνάιντερ σύμβουλος ε, πολιτικής ε, στην ε, Συμβουλευτική Επιτροπή των Συνδικάτων στον ΩΣΑ. Εργάζεται σε δικαιώματα θέματα πολιτικής εργασίας, εκπαίδευσης. Έχετε το λόγο. Καλώς όρισατε. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να, μου δώσει να σας αναφέρω κάποια στοιχεία για την ε, απελευθέρωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Κορέα. Οι οικονομολόγοι ε, πολλές φορές λένε ότι ε, υπάρχει ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εμείς είμαστε μια συμβουλευτική ομάδα και γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται με την Κορέα γιατί έχουμε αρκετά μέλη μας που είναι επιτόπου στην Κορέα και εργάζονται εκεί. Ε, πρόεδρε, έχει υποθεί ότι η ε, συμφωνία αυτή είναι η πιο πλήρης με την ε, Κορέα, η πιο πλήρης συμφωνία ε, ελεύθερων συναλλαγών που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ ενδιαφέρον ως προς αυτό, τουλάχιστον από την πλευρά των συνδικάτων, είναι οι διατάξεις των κεφαλαίων 13 και 15 της συμφωνίας τα οποία θα διευκολύνουν την συμμόρφωση με, τους, ε, με τα πρότυπα του, της ΔΟΕ και με την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία που βεβαίω θα, υπάρχει και θα συνοδεύεται και από ισχυρό σημαντικό ε, μηχανισμό ελέγχου, παρακολούθησης, ε, θα υπάρχει συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών, συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων, συνδικάτων κτλ. Το βασικό ερώτημα για τα συνδικάτα ως προς αυτό είναι το εξή. Μπορούμε να περιμένουμε από τις κορατικές αρχές να είναι σοβαρές και να λάβουν σοβαρά τη δέσμευσή τους ε, για την συμμόρφωση με την αξιοπρεπή εργασία και τα πρότυπα, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 13. Και για να μπορέσει να απαντήσει κανείς το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να λάβει και την ε, υπόψη του και την ε, εμπειρία που υπάρχει με το εργατικό δίκαιο που έχει υπάρξει στην ε, Κορέα, καθώς επίσης και την μεταρρύθμιση που έχει γίνει στη χώρα. Βέβαια τα, η εμπειρία αυτή δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Πριν όμως αναφερθώ στην Κορέα, να σχολιάσω κάποια από, τα βασικά, από τις βασικές διατάξεις του κεφαλαίου 13. Τα συνδικάτα θα έχετε δει ότι επειδή κάποιοι από τους οργανισμούς μας έχουν εκδώσει ανακοινωθέντα τύπου, τα συνδικάτα ε, ε, εκτιμούν τις αναφορές που γίνονται για να συμπεριληφθούν αυτά τα πρότυπα εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία στα, στο 13.4 και στο 13.6 της συμφωνίας, στα σχετικά άρθρα. Η, επίσης ε, αυτό αφορά και την δέσμευση της, εφαρμογής, της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμβάσεων της ΔΟΕ και επίσης καλωσορίζουμε την ε, συμφωνία ότι δηλαδή τα μέρη δεν θα αποδυναμώσουν την, ε, το ρόλο των ε, οργανισμών της αγοράς εργασίας για να ενισχύσουν το εμπόριο. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ, έτσι διαβάζω εγώ αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Τώρα, στη αφορά την Κορέα, η δέσμευση που αφορά την αναγνώριση των εργασιακών προτύπων βρίσκονται σε μεγάλη αντίθεση με τις πολιτικές για το εργατικό δίκαιο και τις βιομηχανικές σχέσεις και τη σχετική μεταρρύθμιση. Η British Weekly και ο Economist ε, αναφέρουν την κατάσταση των συνδικάτων στην Κορέα και εν περιλήψη λένε ποια είναι τα πρώτα πρόσφατα μέτρα που, προτείνουν, ε, που πρότεινε ο πρόεδρος που ε, και υιοθέτησε η συνέλευση των ε, στην Κορέα. Τα μέτρα αυτά έχουν ε, σχεδιαστεί και εφαρμοστεί για να αποδυναμώσουν τα συνδικάτα και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να πω εδώ ότι η κυβέρνηση έχει καταπιέσει τις εργασιακές σχέσεις στην Κορέα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό Ειδικά φαίνεται από το ότι ο υψηλός αριθμός, υψηλός αριθμός συνδικαλιστών έχουν ε, συλληφθεί μόνο και μόνο επειδή κάνουν τα καθήκοντα που τους αρμόζουν, οργανώνουν τους ε, εργαζόμενους για να γίνουν μέλη, προσπαθούν να διαπραγματευτούν ε, τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και σύμφωνα με κάποια στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που υπάρχουν ε, από τι ε, ε, εταιρείε μα στην Κορέα για τα τελευταία 12 χρόνια, και το τονίζω 12 χρόνια, γιατί αυτή η περίοδος καλύπτει τρεις διαφορετικούς, τρεις διαφορετικές θητείες προεδρικές. Τα, τα δεδομένα λοιπόν, οι συλληφθέντες συνδικαλιστές είναι περίπου 2.200 και αν μιλήσουμε με προσώπους της ε, Κορέας την Παρασκευή θα, μας, ε, θα μου θέσουν το ερώτημα ε, πόσοι όμως συνδικαλιστές έχουν συλληφθεί, συλληφθήσαν χτες ας πούμε στη Γαλλία και εγώ αν πω συγγνώμη γιατί πρέπει δηλαδή να συλλαμβάνονται στη Γαλλία οι συνδικαλιστές θα μας πούνε να όμως από χτες έγινε απεργία στις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος πάντων θα επανέλθω σε αυτό ε, αυτό είναι ένα θέμα στην Κορέα, το να κάνει κανεί απεργία. Γιατί ο, τομέας, ο κλάδος των υπηρεσιών δεν συνάδει με τις συστάσεις του, της ΔΟΕ. Οι, ε, τα συνδικάτα λοιπόν έχουν ε, αναφέρει συχνά τις συστάσεις που τους γίνονται από τον ΩΣΑ, αλλά δεν έχουν συμμορφωθεί με την συμφωνία που προκύπτει από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι πρωτογενές δίκαιο και δίνει τη δυνατότητα ε, να, γίνει, να υπάρξει συμμόρφωση αλλά οι Κορεάτες δεν έχουν κάνει τίποτα ακριβό, τίποτα απολύτως για να εφαρμόσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ό,τι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κορέα. Και τέλος, Πρόεδρε, να πω ότι καμία από τις διατάξεις της συμφωνίας, ειδικά στο κεφάλαιο 13, δεν αναφέρεται στην ε, δήλωση της G20 και των εμπειρογνωμόνων. Εδώ όμως το ερώτημα είναι πόσο σοβαροί είναι οι Κορεάτες σχετικά με τη δική τους δέσμευση. Η επόμενη διαφάνεια απλώς αναφέρεται σε μία ε, πρόσφατη έκθεση που εξεδόθη από την, από την ΕΤΟΚ που βρίσκεται εδώ στις Βρυξέλλες και είναι μία έκθεση για την παραβίαση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά θα ήθελα εδώ να μοιραστώ μαζί σας τουλάχιστον έτσι κάποιους τίτλους για, τις, για, την, για το τι έγινε στην Κορέα. Καταρχήν υπάρχει μια συνεχιζόμενη καταπίεση σε ό,τι αφορά την οργάνωση σε συνδικαλιστικά κινήματα συλλήψεις λόγω δραστηριοτήτων συνδικαλιστικών. Αυτό είναι το, το κλασικό που κάνουν. Αν πούμε, κάποιος είναι ακτιβιστής, συνδικαλιστής, αντιμετωπίζει φυλάκιση, δίωξη και αυτό αναφέρεται και στον ποινικό κώδικα του, στην Κορέα που περιγράφει ακριβώς ε, ότι είναι παρακόλληση των, επιχειρη... των δραστηριοτήτων και οι συνδικαλιστές έχουν μηνυθεί πολλές φορές και από επιχειρήσεις και υπάρχουν και άλλα θέματα που προκύπτουν από τον δημόσιο τομέα ας πούμε οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κορέα δεν επιτρέπεται να δρουν σε ό,τι αφορά να δρουν συμμορφούμενοι με τα πρότυπα. Πολλοί, δημοσιοί πάλι δεν μπορούν να, δεν επαγορεύεται να είναι μέλη συνδικαλιστικών κινημάτων και τέλος υπάρχει και το θέμα της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλές φορές απολύονται από τους εργοδότες τους εάν συμμετέχουν σε δράσεις σε συνδικαστικών κινημάτων που θεωρούνται α, ως προσπάθεια να εκφραστεί μια πολιτική αντίθεση στην Κορέα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν στην Κορέα δεν επιτρέπεται να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων, δεν μπορούν να είναι ενεργά μέλη πολιτικών κομμάτων και μια πρόσφατη περίπτωση τέτοια ήταν μια προσπάθεια 134 δασκάλων που δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά μόνο συμμετείχαν σε μια διαδήλωση ενός συνδικάτου που καταδίκαζε τις ε, πολιτικές της κυβέρνησης. Ένα τελευταίο θέμα, Πρόεδρε, έχει να κάνει με την παρέμβαση της κυβέρνησης στα συνδικαλιστικά. Η κορεατική κυβέρνηση δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της ούτε τις συστάσεις της ΔΟΕ, ούτε και τις συστάσεις που προέρχονται από τον έλεγχο και από την όλη διαδικασία που ασκεί ο ΩΣΑ. Θα έχετε ίσως ε, δει, ίσως να το γνωρίζετε, ότι η Κορέα έγινε μέλος του ΩΣΑ το 1996. Αλλά λόγω των ε, πολιτικών ο ΣΑ θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια ειδική ελεγκτική διαδικασία για να χρησιμοποιηθεί αυτή η πίεση ομοτήμων ως εργαλείο για να ε, υποστηριχθεί το εργατικό δίκαιο και η μεταρρύθμιση στην ε, Κορέα. Παρόλα αυτά, και λόγω και του επιτυχούς λόμπι που έκαναν οι, η κυβέρνηση της Κορέας αυτό, αυτή η διαδικασία δεν, ε, δεν πέτυχε τελικά τον βασικό του στόχο. πρόεδρε, ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο να κλείσω απλώς λέγοντας ότι τα συνδικάτα θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να είναι, αν θέλουν να είναι σοβαρά για την αποτελεσματική εφαρμογή και πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με τους Κορεάτες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό που έχουν, τις πίεσεις ομοτήμων, για να πιέσουν τις κορεατικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που υπέγραψαν ε, και που θα τεθούν ενισχύ με την υπογραφή της συμφωνίας. Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν το κάνουν, αυτό θα συμβάλλει στο, στην, ε, στο να δημιουργηθούν προβλήματα σε ό,τι αφορά τι ελεύθερε συναλλαγέ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στις 11 παρα 25. Μας, δεν μας έχουν μείνει 25 λεπτά. Uh, Γι' αυτό θα ήθελα να δείξετε εγκράτεια στη συζήτηση και να μην μακρηγορείτε. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στους συζητητές μας, τον κύριο Ρομπερτ Στέρντι, που είναι ο εισηγητής ε, για την ίδια τη Συμφωνία Ελεύθερα Μπορεί και στον Κρόντιο Φάβερ, που είναι ο εισηγητής για τη ρήτρα της διασφάλισης. Κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στους κυρίους Γουλστοκ και Γινάθιο Καρθία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ενδεχομένω ε, της ομίγυρης. Και παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Τρία λεπτά στον κύριο Στέρντι που είναι και ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Δεν θα τα εξαντλήσω καν αυτά τα τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας για τη συμμετοχή τους εδώ. Ήταν συναρπαστική η παρουσίαση, όλες οι παρουσιάσεις ε, και πολύ παιδαγωγικές. Μάθαμε πάρα πολλά και νομίζω ότι ε, επιβεβαιώθηκε η θέση μας και από τα δικά σας επιχειρήματα. Κύριε Κερνέης, μπορείτε να μου απαντήσετε αργότερα, αλλά αν δεν προλαβαίνετε μπορείτε να μου στείλετε και γραπτός ε, την απάντηση. Όταν ο Κορεάτης Υπουργός Εμπορίου ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρώτησε τι γίνεται με τις υπηρεσίες των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Μου είπε ότι θα συναυθεί ειδική συμφωνία για το θέμα αυτό. Προς το παρόν είναι κλειστή αυτή η αγορά. Ξέρετε αν έχει συναυθεί αυτή η συμφωνία ή ξεκολουθεί αυτός ο κλάδος να είναι κλειστός στην Κορέα. Ο κ. Φάβαρ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ συνοπτικά να διευκρινίσω ότι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα αποφέρει ωφέλη και στην Ευρώπη αλλά και στην ε, Κορέα. Θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική διαπραγμάτευση σίγουρα, αλλά γιατί να μην αξιοποιήσουμε τις θετικές πτυχές αυτής της συμφωνίας. Εγώ είμαι ένθερμο υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, πολύ περισσότερο στην εποχή αυτή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Επίσης, ε, είμαι υπέρμοχος των ισορροπημένων ε, εμπορικών συμφωνιών των ισορροπημένων και για τους δύο εταίρους και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιθανά ωφέλη που θα αποκομίσουν τρίτες χώρες από τη συμφωνία αυτή. Έχω την αίσθηση και περιμένω και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα συνάψουμε και με άλλες χώρες συμφωνία ελεύθερο εμπόριο, όπως με την Κίνα. Γνωρίζουμε ότι το κόστος παραγωγής στην Κίνα είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στη Νότια Κορέα και φυσικά πολύ χαμηλότερο το κόστος αυτό από ό,τι στην Ευρώπη. Και η συμφωνία αυτή θα είναι τελείω ε, άνηση, γιατί εμεί δεν έχουμε σχεδόν καμία πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την άποψη αυτή. Μπορεί να είναι βέβαια εσφαλμένη η προσέγγιση μου. Επίση, ε, έχω και μία ερώτηση προ οποιοδήποτε αρμόδιο. Φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο για νέα ρυθμίση διοξιδίου του άνθρακα στα αυτοκίνητα της Κορέας που πολύ πιθανόν να επηρεάσει και τους ε, Ευρωπαίους αυτοκινητοβιομηχάνους. Έχετε αξιολογήσει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της νέας αυτής ρύθμισης ε, προς τις εξαγωγές μας για στην Κορέα. Ωραία, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Φάρτιν από το ΕΛΚ, μάλλον ο κύριος Κάσιντι. Τρία λεπτά έχετε κι εσείς κύριε Εγώ έχω αρκετές επιφυλάξεις. Έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν για να διασκεδάσω τις ανησυχίες μου. Είπαμε για την χημική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι μη δεσμολογικοί φραγμοί με τη συμφωνία αυτή ελεύθερο εμπόριο. Ακόμη και κάτι που είναι πολύ θετικό για τη χημική βιομηχανία. Έχετε όμως λάβει εχέγγυα από την κορεατική πλευρά για την κατάργηση αυτή. Γιατί βλέπουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, ότι από το 1985 και μετά είχαμε εισαγωγές, με μόνιμη υποχρέωση κατάργησης των μη δεσμολογικών φραγμών. Παρ' όλα αυτά, αντί να έχουμε κατάργηση, είχαμε όλο και ενίσχυσή τους. Και μάλιστα όσοι αγόρασαν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και βλέπουμε τις εκπομπές δεξιδίου του άνθρακα, διαπιστώνουμε τις διαφορές. Πώς θα εξασφαλίσετε επαναφορά των ε, μη δεσμολογικών φραγμών και μάλιστα δρυμύτερων. Επίσης ε, υπάρχει ένας κανόνας στη συμφωνία αυτή. Πώς θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του κανόνα αυτού στην Κορέα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αδίκημα της παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης. Πώς ε, θα εξασφαλίσετε την ε, σωστή εφαρμογή των συμπεφωνηθέντων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διάπραξη αδικημάτων. Ο κύριος Ζαλεύσκη, αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής μας, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έδειξε πόσο πολυσύνθετη είναι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και τι πολυάριθμες ε, επιπτώσεις έχει σε διάφορους κλάδους. Για παράδειγμα για, την, ε, για τον κλάδο των υπηρεσιών είναι υποφελής αυτή η συμφωνία. Και έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα επιδράσει τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η συμφωνία αυτή. Βέβαια υπάρχουν και πολέμοι επικριτές αυτής της συμφωνίας. Για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μάλλον ενάντια της συμφωνίας αυτής, έχει σοβαρές επιφυλάξεις για τη σύναψή τη. Οπότε εμείς θα πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθεί και να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε να τονώσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή οικονομία ή γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία είναι τεχνολογία υψηλή και η καινοτομία συγκεντρώνεται στους ισχυρότερους. Οπότε διαρωτώ θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε σε μακροπρόθεσμη προοπτική τον ηγετικό μας ρόλο ε, στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, σε περίπτωση που ανοίξουμε την ευρωπαϊκή αγορά στους κορεατικούς παραγωγούς θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε αυτή την ηγετική θέση τη Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία και μετά τη σύναψη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση πριν προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και κύρωση αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Περιμένω λοιπόν απαντήσει από του καλεσμένου. Τώρα από εδώ και πέρα δύο λεπτά θα δικαιούται ο κάθε ομιλητή. Από τους φιλελεύθερους, ε, τους πράσινους, ίσως ο κύριος Με Μένω ε, με ορισμένες αξιολογήσεις για τα ωφέλη μιας τέτοιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Καταρχήν οι μελέτες επιπτώσεων επικεντρώνονται στα μελλοντικά ωφέλη. Δεν γίνονται ποτέ μελέτες επιπτώσεων για την εφαρμογή, για την πραγματικότητα, για το παρόν ε, τέτοιων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και πώς επηρεάζουν τις οικονομίες μας σήμερα. Για παράδειγμα, εγώ εκλέγομαι από τη Δυτική Γαλλία και μου λένε πολύ ωραία η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε χείρου στην Κορέα. Στη Δυτική Γαλλία ίσω εκεί ο τζίρο ε, τη επιστημιστική βιομηχανία για το χείριο κρέατο είναι υψηλό. Αλλά εκεί θα έχουμε μείωση απασχόλησης τη εντατικοποίηση τη παραγωγή. ένα τμήμα του πληθυσμού θα χρειαστεί να αγοράσει εφιαλωμένο νερό, γιατί υπάρχει μόλυνση των πηγών. Επίσης ε, υπάρχει πρόβλημα του τουρισμού στη Βρετάνη εξαιτίας ε, του πολλαπλασιασμού των πράσινων φυκιών. Ε, ή υπάρχει ένας τομέας που ζει από την παραγωγή σόγιας της Λατινικής Αμερικής που όμως τροφοδοτείται από την αποψήλωση των δασών της Αμαζονίας. Βλέπετε τις διάφορες επιπτώσεις λοιπόν. Επίσης άκουσα την αυτοκινητομηχανία να ζητά την προστασία μας. Τι έγινε ε, Ποιο ήταν ο τζίρο τη αυτοκινητοβιομηχανία του τελευταίου μήνε, 40-50 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε όμω η αυτοκινητοβιομηχανία από τη στήριξη των 40-50 δισεκατομμυρίων ευρώ που έλαβε από τι κυβερνήσει. Τα χρησιμοποίησε για να επιμορφώσει, να ανακυκλώσει του εργαζόμενου τη ή να κάνει πιο καινοτόμα αυτοκίνητα, ε, να παραγάγει πιο μικρά αυτοκίνητα, λιγότερο ρηπαίνοντα και πιο προσαρμοσμένα στις συνθήκες των πόλεων. Τι έκανε λοιπόν η αυτοκινητοβιομηχανία, μόνο προστασία ζητάει και μάλιστα όπως και η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό στη στάση της. Ναι, να προστατεύσουμε μια αυτοκινητοβιομηχανία που δεσμεύεται να, να να εγκληματιστεί στις νέες συνθήκες και στην κοινωνία και στις παγκόσμιες συνθήκες, όχι όμως μόνο για να επωφεληθεί από κάποιες εξαιρέσεις στην κορεατική αγορά και να μην τηρήσει τους, τις νέες ρυθμίσεις και τους αυστηρότερους κανόνες για το διοξείδιο του άνθρακα, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Δύο σχόλια μόνο. Και εγώ θα ήθελα να πω κάτι για την αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ δεν με ρολυπτώ, γιατί κατάγομαι από μια χώρα που εμπορεύονται και εμπορικά αυτοκίνητα αλλά και κορεατικά. Οπότε προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, δεν έχω προκαταλήψει υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Πάντως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά το θέμα των νέων φραγμών, των μη δασμολογικών φραγμών και το θέμα της ε, επιστροφής των δασμών, του duty drawback. Υπάρχουν άλλες ε, εναλλακτικέ λύσεις για αυτά τα δύο θέματα, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ε, στον εκπρόσωπο του ΣΕΦΙΚ, θα υπάρξουν κάποια μέτρα ε, με βάση τη Συμφωνία Ρίτς για τις αγωγές χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να, να γίνουν κάποιες επιπτώσεις, να γίνει μια σύγκριση εισαγωγών-εξαγωγών χημικών προϊόντων και στο εσωτερικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάραντελ ο Τζο Χίγγινς από την ΚΟΕ. Δύο λεπτά κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Κανονικά σε τέτοιες ακροάσεις, πρόεδρε, υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, διαμάχες ανάμεσα στο κεφάλαιο και τα συνδικάτα. Αυτή τη φορά το κεφάλαιο ενωμένο μιλάει για τα ωφέλη από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την ε, Κορέα. Εμείς διαφωνούμε με την αυτοκινητοβιομηχανία από την μια μεριά και ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να περιμένει τι θα γίνει με τις ιδιωτικοποίησεις. Αυτό λοιπόν που εγώ θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή είναι λιγάκι να παίξει το διαιτητή εδώ. 20.000 θέσεις απασχόλησης που ακούμε ότι θα χαθούν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι και αυτό κομμάτι της αξιολόγησής σας. Και ποιο είναι το συμπέρασμα για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Ο χημικός τομέας, οι υπηρεσίες πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ καλή για αυτούς. Ναι, αλλά για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει την απάντηση. Και ποιες είναι οι συνέπειες της ε, μετακίνησης εργατικού δυναμικού εδώ. Επίσης, Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα την Επιτροπή. Η έκθεση που ακούσαμε από τα συνδικάτα και από ό,τι ξέρουμε και από δικές μας εκθέσεις, είναι πράγματα πολύ ανησυχητικά. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μας λέει για τη συμμόρφωση της Κορέας στις διατάξεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό στα λόγια. Στην πραγματικότητα όμως, τι θα αλλάξει για τους Κορεάτες εργαζόμενους, για τα δικά τους τα δικαιώματα, εφόσον υπογραφεί, επικυρωθεί η συμφωνία αυτή. Θέλω να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, από την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας, κανείς. Από τους υπόλοιπους έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Γιάννουσαν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ πέρα κάναμε κάποιο λάθος. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπέρ της ελεύθερης, ε, ε, ελεύθερη, συναλλαγών και από την άλλη μεριά υπέρ του προτεξιονισμού, του προστατευτισμού, ε, κάνουμε λάθος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που καταπιέζει τη ελευθερία του άλλου. Οπότε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Αναφέρεται και στα ανακοινωθέν τύπου λιγάκι αυτά. Λοιπόν, εγώ συγκράτησα το εμπορικό έλλειμμα που θα είναι στα 5 δισεκατομμύρια για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα κερδίσουμε όμως τις υπηρεσίες. Έχουμε και τη χημεία που θα έχει πλεόνεσμα 1,5 Ωραία, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όμως ένα δεδομένο. Η μεγάλη ευκολία με την οποία προχωράνε οι μετεγκαταστάσεις των υπηρεσιών, όχι μόνο των βιομηχανιών. Και το άλλο είναι ότι είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να δώσουμε ζωντάνια στην αγορά των υπηρεσιών παρά της βιομηχανίας. Μα αφήστε με να μιλήσω ένα μισή λεπτό πρόεδρε, μην με κόβετε. Λέω Λοιπόν, υπάρχει μια προσέγγιση εδώ, η οποία λείπει πιστεύω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, ωραία. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, οπότε ας ακούσουμε τον καθηγητή Βίλκοκ και τον ε, κύριο Γκαρθία. Οκτώ λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, τέσσερα λεπτά ο καθένας λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά Βίλκοκ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω εγώ σε δύο ερωτήσεις και οι συνάδελφοί μου σε άλλε δύο. Για το θέμα αυτό της διασφάλισης ότι δεν θα υπάρχουν τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια εγγύηση σε οποιαδήποτε αμοιβαία συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσει να μην υιοθετήσει τίποτα νέε ρυθμίσει. Άπαξ και το κάνει αυτό και το κάνει συνεχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαν να παραβαίνει αυτή τη συμφωνία. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εγγύηση. Μπορείτε να πάτε όσο γίνεται πιο μακριά για να διασφαλίσετε ότι οι τεχνικές ρυθμίσεις δεν στρεβλώνουν το εμπόριο, ναι. Πάντως η συμφωνία αυτή πάει πιο μακριά από ό,τι έχουμε πετύχει στον ΠΟΕ ποτέ μέχρι τώρα. Τώρα για τις συνέπειες. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Αν δούμε τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα, αξιολογούμε ότι οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι μικρές. Όντως θα υπάρξουν κάποιες μετεγκαταστάσεις, αναγκαία, είναι αναπόφευκτο. Σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία το έχουμε αυτό. Πάντως από τα στοιχεία που έχουμε για την απώλεια θέσεων απασχόληση στην αυτοκινητοβιομηχανία, Συγχρόνω έχουμε εξαιτία των επενδύσεων των Κορεατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια αύξηση. Ένα τομέα πάντως που δεν αναφέρθηκε σήμερα το πρωί είναι η μηχανική που έχει ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Δεν το αναφέραμε σήμερα το πρωί. Αυτά από τη δικιά μου την πλευρά και μήπως ο Τζακ έχει κάτι να προσθέσει εδώ. Παρακαλώ. Για τις επιστροφές δασμών, το duty drawback. Η μελέτη που δώσαμε στην ε, Επιτροπή σας έχει ένα μεγάλο παράρτημα ακριβώς για αυτό το θέμα. Μπορούμε πάνω από τα χίλια ευρώ για τα αυτοκίνητα να έχουμε ένα 320. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό αλλά υπάρχουν πολλά σενάρια ανάλογα με το ποσοστό των εισαγωγών τώρα στο μέλλον. Φτάνουμε στα 3,20. Αλλά πιο πολύ είναι της τάξης του 100 ή κάτι τέτοιο. Και ναι, δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν το αρνούμε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αρνείται, αλλά οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες. Και αν θέλετε να φτάσετε στα σενάρια τα πιο ακραία, θα βρείτε τις λεπτομέρειες στο παράρτημα που σας έχουμε δώσει. Πρόεδρος, ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο Ιγνάθιο Γκαρθία. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Καταρχήν για το εμπορικό ισοζύγιο. Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ακριβώς το ισοζύγιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κορέα που καταλήγει σε πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάξω στο 10 δις που σημαίνει μεγάλη μείωση του ελλείμματος που είχαμε μέχρι τώρα στο ισοζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν δείτε τι έγινε μετά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΦΤΑ τι ΕΖΕΣ, των χωρό ΕΖΕΣ δηλαδή με την Κορέα, θα δείτε ότι τότε είχαμε αύξηση του 5%. Αν δείτε το συνολικό ισολογισμό, έχουμε ένα αποτέλεσμα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να αυξηθεί το έλλειμμα. Αλλά το είπε ο κύριος ο καθηγητής Βίλκοκ ότι η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα χάρη στις επενδύσεις της Κορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τρίτες χώρες. Θα δείτε ότι οι εξαγωγές από την Κορέα έχουν μειωθεί, ενώ οι πωλήσει των κορεατικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί. Για το... Συγχρόνως εμείς πιστεύουμε, με μετά από αυτά που είπε και ο καθηγητής Βίλκοκ, ότι Όντω οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι μικρές και ό,τι προβλήματα υπάρχουν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον μηχανισμό που έχουμε προβλέψει από το Ταμείο για τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση. Τώρα για τις επιστροφές δασμό, το duty drawback. Όντως υπάρχει ένα παράρτημα του LC όπου θα τα βρείτε όλα. Συμφωνώ με όσα αναφέρει το παράτημα και σας ενθαρρύνω να το μελετήσετε. Αυτό πάντως που βγαίνει ξεκάθαρα είναι ότι οι επιπτώσει θα είναι τη τάξη του 1% τη αξία του αυτοκινήτου και στην χειρότερη περίπτωση μπορεί να φτάσει στο 2% τη αξία του οχήματο. Αυτά για την οικονομική διάσταση των επιστροφών δασμών. Έχουμε επίσης κρατήσει τους κανόνες καταγωγής για όλους τους ευαίσθητους τομείς Είναι μια συμφωνία λοιπόν από την οποία εποφελούνται οι τρίτες χώρες, αλλά εμείς κρατάμε για τους ευαίσθητους τομείς τη διάταξη αυτή. Τώρα για, τις μη, για τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Όντως, προσπαθήσαμε στην αυτοκίνητοβιομηχανία να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον, την άλλη πλευρά να ρυθμίσει και η Κορέα έχει δικαίωμα να ρυθμίσει για το περιβάλλον και εμείς έχουμε δικαίωμα να ρυθμίσουμε για το περιβάλλον. Αν δείτε, οι περιορισμοί πάντως είναι πολύ λίγοι όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Οι διατάξεις αυτές είναι δεσμευτικές. Πάντως, Μπορώ να σας καθισχάσω κύριε Χόντακο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Άπαξ και κάποιο ρυθμιστικό μέτρο εντοπίζεται ως ε, μέτρο το οποίο πλήττει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, αμέσως θα παρέμβουμε. Είναι κάτι που το κάνουμε έτσι κι αλλιώς με το διοξίδιο του άνθρακα σε στενή συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία και θα φροντίσουμε να υπάρχει ισορροπία. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την Κορέα να ρυθμίσει για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η ρύθμιση αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πλήττει τη δικιά μας πρόσβαση στην αγορά τους. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και το τι γίνεται στην Κορέα. Εμείς χρησιμοποιούμε ό,τι δυνατότητες έχουμε ε, από τη συμφωνία αυτή σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα για να πιέσουμε την Κορέα να βελτιώσει τις πρακτικές της. Και ξέρω ότι ο κύριος Γιονγμόν που ε, είναι η υπουργό, είπε ότι στηρίζει τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε λοιπόν την ακρόαση πολύ επικοδομητική. Ακούσαμε τις απόψεις τριών από τα μεγαλύτερα μέρη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ακούσαμε τους εργαζόμενους, ακούσαμε ανεξάρτητο ε, εμπειρογνώμονα, ακούσαμε και την Κομισιόν. Οι συζητήσεις μας θα συνεχιστούν βέβαια, τουλάχιστον για την συμφωνία αυτή καθ' αυτή σε λίγο θα κάνουμε την ψηφοφορία για τον κανονισμό για την διασφάλιση. Ευχαριστώ λοιπόν όλους που συμμετείχαν στην ακρόαση και για την συμβολή σας.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλώ να σταματήσω τα πηγαδάκια. αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Ψηφοφορία για τη δημερή ρήτρα διασφάλισης στην Συμφωνία Ελεύθερη Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας. Έχουμε, έχουν κατατεθεί 130 τροπολογίες, αλλά ο εισηγητής και οι σκιώδεις ε, εισηγητές κατάφεραν και συνεννοήθηκαν να τις περιορίσουν σε 14 συμβαστικές τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία και θα ήθελα να σας θερμοπαρακαλέσω να κάνετε ησυχία όσο γίνεται. Καθίστε παρακαλώ. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 44, 45, 46 και 47 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 54, 55, 56 και 58 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ε, Compromise amendment number two. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Against. Abstentions. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 66, 67 και 64W είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 5. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε χωριστά. Ο κύριος Ζάλμπα. Έχουμε και προφορική τροπολογία. Το ΜΕΙ δύναται, αντικαθίστε το ΣΟΥΝΤ ε, θα όφιλε. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 5. Α, ο λάθο λέει ο κύριο Άλμπα. Λάθος δικό μου λέει ο κύριο Άλμπα. Για το τοπικό, τη τοπική συμβουλευτική ομάδα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 77 και 78 παρόμοιε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 80. κατά αποχές εγκρίνεται. 79 και 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 και 82. Ή μάλλον όχι μόνο 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 ποιος είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ της 90 κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 7 ποιος είναι υπέρ ο Παύλος Ζάλβα τώρα είναι που θα ήθελα να προσθέσουμε την προφορική τροπολογία και το May να αντικατασταθεί από το should. Στη συμβαστική τροπολογία 7 υπάρχουν αντιρρήσεις με την προφορική τροπολογία, αντικατάσταση του δύναται από το θαόφιλε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 7 με την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 95 και 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 95 και 98. Άρχιτη ψηφοφορία. And the vote is... Τέλος ψηφοφορίας. Everyone. So please make up your minds. Αποφασίστε επιτέλους. Τώρα τέλος ψηφοφορίας. Μ, ισοπαλία. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 του Μπέντ Λάγκε. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ποιες Εγκρίνεται. 97. ποιο είναι υπέρ. Κατά. όχι. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Την παραγραφό 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα είναι η παράγραφος 3. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον καταπίπτει γιατί κατηλείπτεται από τη συμβαστική λύση. Οπότε περάμε στην τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογίες 104 και 105. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 107. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Τροπολογία 112 119 και 122 ψηφίζουμε πρώτα την 112 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε θα ψηφίσουμε χωριστά τις άλλες. Την παράγραφο 2 μόνο, ξεχωριστά. Νομίζω όμως ότι είχε απορριφθεί. Α. 113 δεν ψηφίζουμε για χωριστά και 130 μαζί ποιος είναι υπέρ 113 και 130 παρακαλώ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 114 και 127 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές 115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 και 128. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τέσσερις παραμεστροπολογίες. 117, 118, 124, 129. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 26D, D, δέλτα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 δ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 ποιος είναι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 11 ποιος είναι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 12 περ κατά αποχές εγκρίνεται 31 ποιος είναι υπέρ κατά Επαναλαμβάνω. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 31. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 2 του Μπέντ Λάγκε υπάρχουν αντιρρήσεις μήπως με την προφορική τροπολογία όχι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογικές σκέψεις, ε, τροπολογίες... Τροπολογία 39, ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 40 άρτη ψηφοφορία τέλος εγκρινήθηκε τροπολογία 42 ποιος είναι υπέρ κατά και πάλι 42 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 43. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίζουμε την ούτως τροποποιηθήσα πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πανψηφί με μία αποχή εγκρίνεται. Έχουμε όμως και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ομοφωνία και πάλι. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά, συγχαρητήρια και στους Κιώδης. Thank you very much. Uh, it's uh, point, point uh, uh, you can tell her. Ένα λεπτό για να μπορέσουμε να συγχαρούμε τον εισηγητή με την ησυχία μας. de, de... Yes. Yesterday we... Please... Πρόεδρος, παρακαλώ ησυχία. I have your attention, please. Τι απίθαρχοι που είσαστε, λέει ο πρόεδρος. Αν δεν ησυχάσετε, θα υποχρεωθώ να σας ζητήσω να βγείτε από την αίθουσα. Λοιπόν, χτες αναβάλαμε το θέμα των εκθέσεων που είχαν να κάνουν, μάλλον τις εκθέσεις που είχαν να κάνουν με την αντιπροσωπεία μας στην Ιταλία. Το θέμα αυτό. Τώρα λοιπόν, επειδή δουλέψαμε τόσο γρήγορα, έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στη συνάδελφό μας, τη Χριστιάνα Μουσκαρδίνη, για να μας ενημερώσει για την μετάβαση αντιπροσωπείας στην Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία μας πήγε στην Ιταλία 25 με 27 Μαΐου και στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Ζάλβα, ο Ζούτσαν, ο Βίλχριτ και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας λοιπόν πήγε σε δύο ε, περιοχές στη Λομβαρδία και στο Πιεμόντε. Συζητήσαμε εκεί με επιχειρήσεις, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως συζητήσαμε για τις εκθέσεις ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα για παράδειγμα και άλλες εκθέσεις που είναι ζωτική σημασίας για την Επιτροπή μας. Μόλις ψηφίσαμε για τη Συμφωνία για την Κορέα. Επίσης το άλλο μας θέμα ήταν ε, η καταγωγή, η ρήτρα καταγωγής που είναι επίσης ένα θέμα σημαντικό για μας. Στις συναντήσεις που είχαμε με τους υπεύθυνου από την Fiat στο Μαρσάνο, στο ερευνητικό κέντρο εκεί, μιλήσαμε και για τις μελλοντικές επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αναφερθήκαμε επίσης στα περιβαλλοντικά ζητήματα, την αηφόρο ανάπτυξη και τα υβριδικά οχήματα. Όσον αφορά μάλιστα τη συμφωνία ε, με την Κορέα, όπως υπενθυμίσαμε και σήμερα το πρωί. θίξαμε τα πιο επίμαχα ζητήματα. Επίσης συναντηθήκαμε με τη, το πρόεδρο της Κομφιντούνστρια, τον κύριο Τσοκόν επίσης Γενικό Γραμματέα των Συνδικάτων και την κυρία Μαριέρα Φεντέλη. Όλοι αυτοί εκπροσωπούν μέλη της εφαντουργίας. Συζητήσαμε κυρίως για το δεσμευτικό μέτρο της καταγωγής και τι γίνεται με τον ανταγωνισμό προκειμένου ο καταναλωτής να παραμένει ενήμερος για την προέλευση. Επίσης, στήσαμε τα θέματα υγιεινής όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία, δηλαδή υφάσματα που χρωματίζονται με τη διαδικασία του φλού. Ίσως να τα έχετε ακούσει αυτά για την Ιταλία. Κατασχέθηκαν ένα σωρό ρούχα και, αυτό, και παπούτσια από την Κίνα. Μιλήσαμε με εκπροσώπους επίσης της μεταλλουργίας, της χαλιβουργίας και θα θυμόσαστε ότι είχαμε και μια ακρόαση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Χαλιβουργίας πριν από μερικές εβδομάδες. Στην Ιταλία λοιπόν συναντηθήκαμε εκπροσώπους της Ντάλνιμαν, με την EMF που είναι η πιο σημαντική στον κόσμο και πήγαμε και στην ομάδα Τενάρης, στην εταιρεία Τενάρης, τον γκρουπ αυτό όπου διαπιστώσαμε τον τρόπο παραγωγής. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν με τους διαγωνισμούς όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Κυρίως για τις σχέσεις μας με την Τουρκία σε αυτό το τομέα. Στη συνέχεια πήγαμε και επισκεφθήκαμε εργοστάσια αποδηματοποίησης μας εξήγησαν πώς έχει επηρεαστεί η αγορά από τις εισαγωγές, τις κινέζικες, οι οποίοι εισάγουν παπούτσια τα οποία δεν είναι σωστά φτιαγμένα. Ρωσέτη κλπ. τις διάφορες επαφές που είχαμε συναντηθήκαμε και με τον Δήμαρχο του Λίνα, τον πρόεδρο της ε, επαρχίας του Μιλάνου, που μάλιστα ήταν ευρωβουλευτής εδώ στην προηγούμενη θητεία. Συναντηθήκαμε επίσης και με τον Ουπιγάντο, που είναι μια οργάνωση όπου συμμετέχουν οι παραγωγοί ε, προϊόντων όπως είναι οι βίδες, τα μπουλόνια και μιλήσαμε για ζητήματα ασφάλειας προϊόντων που μας έρχονται από τρίτες χώρες. Τέλος, συναντηθήκαμε με τους υπεύθυνους της Λένη που είναι το Εθνικό Όργανο Ηλεκτρισμού, η επιχείρηση δημόσιου ηλεκτρισμού. Όπως ε, και συζητήσαμε θέματα που έχουν να κάνουν με ηλεκτρισμό, με το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Με εκπροσώπους της ΕΝΗ συζητήσαμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία που πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες. Έτσι κάπως σύντομα λοιπόν Αυτά συνέβησαν κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ιταλία. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά θέλω να αποφελθώ από την ευκαιρία εδώ για να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι και που διασφάλισαν την ε, επιτυχία της επίσκεψής μας αυτής. Μας πρότειναν ερωτήσεις για παράδειγμα προκειμένου να συζητήσουμε με τον Ιταλικό βιομηχανικό κόσμο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της, από που πήγαν στην Ιταλία. Ο Παύλο, ο συνάδελφος Σούστα είναι εδώ. Ε, δεν ξέρω αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μουσκαρδίνη και να τη συγχαρώ για την επίσκεψη αυτή. Όντως, πήγαμε στη Fiat και είδαμε από κοντά άμεσα την προβληματική που συνδυάζεται με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μας. Εμένα με βοήθησε η επίσκεψη αυτή, έμαθα πολλά και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή βοήθησε να ολοκληρωθεί με επιτυχία και η εξέταση της ε, έκθεσής μου. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι όλα υπόθηκαν. Τα από όλα, κυρία Μουσκαρδίνη. Ήταν πραγματικά μια επίσκεψη πολύ καλά προετοιμασμένη. Είχαμε επαφές, πρακτικές, πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ήταν επιτυχής η επίσκεψη αυτή και ευτυχώ, πρώτη στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκής ε, Ένωση και δείχνει πόσο επικοδομητικό είναι να κάνουμε τέτοιου είδου επισκέψει. Η επόμενη επίσκεψή μας θα γίνει στην Ουγγαρία. Έτσι λέει το πρόγραμμα, ελπίζω να είναι και αυτή εξίσου επιτυχής και ευχαριστούμε ιδιαίτερως την Κριστιάνα Μοσκαρντίνη για τη δουλειά που έκανε προεδρεύουσα αυτή της επιτροπή. Λοιπόν, να κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα γιατί περιμένουμε την ε, ε, προσκεκλημένη μας από την ε, Ισπανική κυβέρνηση. Για να ακούσουμε την άποψη της Ισπανικής κυβέρνησης για την πολιτική για το εμπόριο. Well, uh, Ώρα να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και καλωσορίζω εδώ την κυρία Σίλβια Ιράνθο που είναι υφυπουργό εμπορίου της Ισπανικής κυβέρνησης. Θα μας μιλήσει για τον ε, απολογισμό της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά τη διεθνή εμπορική πολιτική. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίζω και τον κύριο Άλφρεντ Βανέτ που είναι εξ αριστερών της και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ λοιπόν. Ήταν μια εξαντλητική συνεδρίαση σήμερα στην Επιτροπή μας και να ξέρετε ότι έχουμε ψηφίσει και τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κορέα. Είναι καλά νέα αυτά. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και άλλες εξηγήσεις, σας δίνω και το λόγο, Σίλβια. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε πρόεδρε και μέλη τη Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από έξι μήνε εντατική εργασία, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνεται ευκαιρία να έρθω και να σα μιλήσω για τα αποτελέσματα τη Ισπανική Προεδρία στον τομέα του Διεθνού Εμπορίου. Όταν ήρθε στην Επιτροπή σα αυτή ο υπουργό Μιγγέλ Σεμπαστιάν τον Ιανουάριο που μα πέρασε, μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας. Και αυτό γιατί καταλαβαίναμε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να αποφεληθούμε από το εξάμεινο αυτό για να δώσουμε νέα όθηση στις θεσμικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα εργαστήκαμε κιόλα. Όπω γνωρίζετε, η Προεδρία δεν έχει εκτελεστικέ αρμοδιότητε, ούτε παίρνει αποφάσει, όμω παίζει ένα ρόλο κλειδί προκειμένου να προγραμματίζονται όλε οι εργασίε γύρω από το Συμβούλιο για μας. Αυτό έχει να κάνει με τις επιτροπές, τις σχετικές με το εμπόριο. Έχουμε έργο συντονιστικό, ε, διευθύνουμε τις εργασίες και φροντίζουμε να δίνουμε όθηση στο έργο μας. Και αυτό ακριβώς κάναμε αυτό το εξάμεινο. Ο απολογισμός της Προεδρίας μας έχει να κάνει κυρίως με το θεσμικό και οικονομικό τομέα. Ξέρετε ότι άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και ότι είχαμε επίσης μία οικονομική κρίση παγκοσμίου ελληνικού. Από τη μια μεριά λοιπόν η Προεδρία μας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τεράστιων θεσμικών αλλαγών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλάβαμε με υπευθυνότητα να προχωρήσουμε στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, φροντίζοντας για την υιοθέτηση αποφάσεων βάσει της νέας λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεχιστούν και τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό κυρίως στον εμπορικό τομέα. Η συνθήκη της Λισαβόνας όντως περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες που έχουν επιπτώσει σε πάρα πολλούς τομείς. Άρα χρειαζόταν ανάλυση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτό ήταν και η προτεραιότητά μας. Εγώ ίδια είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις για το θέμα αυτό στο Στρασβούργο τον ε, Φεβρουάριο με τον Πρόεδρό σας τον κύριο Μορέιρα και με εκπροσώπους από την κάθε πολιτική ομάδα και μπόρεσα να διαπιστώσω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Καρπός της εντατικής αυτής δουλειάς που κάναμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με τα κράτη-μέλη συζητήσαμε για πρόταση κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις που πρέπει να εγκρίνει και το δικό σας σώμα. Μετά από διάφορε συζητήσει που έγιναν για αυτό το θέμα, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τι επόμενε μέρε την ανακοίνωσή τη σχετικά με την μελλοντική πολιτική όσον αφορά τι άμεσε επενδύσει και μια πρόταση κανονισμού για τι διμερεί συμφωνίε επενδύσεων. Επίσης, προωθούμε και τις διαδικασίες έγκρισης της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, Ελεύθερων Συναλλαγών με την Νότια Κορέα και τον εσωτερικό κανονισμό που πρέπει να εγκρίνουμε με συναπόφαση. Από την άλλη πλευρά, πέρα από τις άτυπες επαφές ε, που είχαμε και που σας ανέφερα πριν, ή που ο πρόεδρος Μορέρα είχε με τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας ξεκινήσαμε να διερευνούμε και τις βάσεις για συνεργασία και για τις διαδικασίες προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις από τα τρία θεσμικά όργανα. Το πλαίσιο τώρα της οικονομικής κρίσης μέσα στο οποίο κινηθήκαμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού έβαλε το διεθνές εμπόριο σε αξιοσημείωτη θέση όσον αφορά την επικαιρότητα. Στις συζητήσεις που είχαμε συμφωνήσαμε για την αναγκαιότητα που υπάρχει να ενισχύσουμε τη συνεισφορά που έχει το διεθνέ εμπόριο για να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε ευημερία και απασχόληση. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εξαμήνου Διαπιστώσαμε ευτυχώ ότι δεν υπήρξε κλιμάκωση του προστατευτισμού. Αυτό οφείλεται στην οριμότητα που έδειξαν ε, οι κυβερνήσει κατά τη διάρκεια τη κρίση, αλλά επίση και εξαιτία τη συγκράτηση που διαπιστώσαμε χάρη στου κανόνε του συστήματο πολυμερού εμπορίου. Από τα στοιχεία του ΠΟΕ ξέρουμε ότι έχουμε μια αύξηση του διεθνούς εμπορίου εμπορευμάτων κατά 25% στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι εμπορικέ ροέ ήταν ικανοποιητικέ. Αυτό το δείχνει επίση και η εκτίμηση που έχουμε για μια αύξηση 9,5% για το σύνολο του 2010. Από πλευρά τη ισπανική προεδρία συνεργαστήκαμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Υπουργοί Εμπορίου. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε άτυπα τον Φεβρουάριο, υπό την δικιά μου Προεδρία μάλιστα, για να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση της στρατηγικής 2020 όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ίδιο έκαναν και τα μέλη της Πολιτικής Εμπορικής Επιτροπής στη συνεδρίασή του τον Μάιο. Με το χείρημα αυτό προχωράμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία διαβούλευση δημόσια από τις 2 Ιουνίου όσον αφορά τη μεροντική πολιτική της, ε, του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτή θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλές απαντήσεις από τις διάφορες πλευρέ της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαβούλευση αυτή, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη αξία και νομιμότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Το σύνθημα τη Προεδρίας μα στον τομέα του εμπορίου είναι περισσότερε εμπορικέ ευκαιρίε με λιγότερου φραγμού. Είναι κάτι το οποίο οδήγησε σε πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές από αυτές ή την παγίωση άλλων, όπως επίσης και την ολοκλήρωση μερικών ή το ξεκίνημα νέων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ νέες ευκαιρίες εμπορίου που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς μέσω του ανοίγματο των εξωτερικών αγορών, μέσα βέβαια από σαφείς και συγκεκριμένους κανόνες που όλοι θα τηρούμε. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας όσον αφορά πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ισπανική Προεδρία... Ως... Θεωρεί ως ε, θεμελιώδη άξονα της πολιτικής την πολυμερή διάσταση. Οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απαραίτητε για να διαπιστωθεί η επικοδομητική μα τάση και να τροφοδοτηθεί ο διάλογος και η συζήτηση. Ένας απολογισμό και μια προσπάθεια εξέβρεση ισορροπίας που έγινε για το γύρο της Ντόχα την περασμένη εβδομάδα 22 Μαρτίου στη Γενέβη Δυστυχώ δεν έδωσε την αναμενόμενη όθηση προς τι διαπραγματεύσεις παρόλο που αργότερα έγιναν συναντήσει όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη διαμόρφωση μιας συνένεσης που όμως δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Ευελπιστούμε όμως ότι θα τελεσφορήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τις αβεβαιότητες που βιώσαμε, οι διαπραγματεύσεις της Δόχα εξακολουθούν να είναι ζωντανές, εν αναμονή των πολιτικών συνθήκων και προϋποθέσεων, προκειμένου να περάσουμε στην τελευταία και οριστική φάση διεκπαιρέωσης των διαπραγματεύσεων της Δόχας. Το πρόγραμμα το διμερές και το περιφερειακό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν όπως ξέρετε πολύ φιλόδοξο και μάλιστα η, Ισπανική Προεδρία υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχε θεσπίσει. Σε ό,τι αφορά την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική διαπιστώσαμε τα μεγάλα επιτέγματα της ε, Ισπανικής Προεδρίας σε εμπορικά ζητήματα. Η διάσκεψη κορυφής της Μαδρίτης στις 18 Μαΐου εξήγηλε την σύναψη διαπραγματεύσεων σημαντικών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με Κολομβία και Περού και σύνδεση με την Κεντρική Αμερική. Οι διαπραγματεύσει με το Περού και την Κολομβία είχαν ήδη διεκπαιρεωθεί το Μάρτιο ως προκαταρκτική φάση μιας ευρύτερης συμφωνίας σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινότητα των Άνδρων. Και μάλιστα γίνονται τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να επανέλθει και το Εκουαδόρ στι διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεση με τι χώρε τη Κεντρική Αμερική, αυτή περιλαμβάνει μια ευρεία και βαθιά εμπορική συμφωνία με μια ουσιαστική απελευθέρωση του εμπορίου των προϊόντων και μια φιλόδοξη κάλυψη των υπηρεσιών, των δημοσίων προμηθειών, των επενδύσεων και της πνευματικής ιδιοκτησία. Έτσι θα προωθήσουμε μια μεγαλύτερη εμπορική ολοκλήρωση στην περιοχή και είμαι βέβαια ότι από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες αυτές μετά τις διαδικασίες ε, έγκρισης που έχουν ξεκινήσει, θα δώσουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας και θα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και των εμπορικών μας εταίρων. Από την, την άλλη πλευρά, η συνέχιση των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερικοσούρ αποφασίστηκε στις 4 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια σειρά τύπων συνομιλιών όπου προσδιορίστηκε ότι τα επίπεδα φιλοδοξίας και των δύο συμβολωμένων μερών επιτρέπουν την ε, επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είχαν διακοπεί για μία πενταετία. Συνεχίζονται όμως για τη δημιουργία μιας ε, πολύ σημαντικής ε, διαπεριφερειακής εμπορικής συμφωνίας με πάνω από 700 εκατομμύρια κατοίκους. Βέβαια θα είναι δυσχερείς οι διαπραγματεύσεις, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθούν σχετικά σύντομα. Η πρώτη, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα γίνει στον Buenos Aires την επόμενη εβδομάδα και εκεί θα δούμε τις συγκεκριμένες θέσεις και προσεγγίσεις για τα επιμέρους κεφάλαια. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία της Βαρκελόνης και την Ένωση για τη Μεσόγειο, εκεί προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την οικονομική ολοκλήρωση και να προωθήσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια και ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα η διοργάνωση τη Γρανάδα το Μάρτιο της πρώτης διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου ε, έδωσε την αφετηρία για μια στενότερη σχέση με τη χώρα αυτή στα πλαίσια του ενισχυμένου καθεστώτος. Ελπίζουμε ότι θα υλοποιήσουμε το στόχο μιας ευρύτερης ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την άποψη αυτή την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση για την ε, για την ίδρυση της ε, γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο στη Βαρκελόνη. Έγιναν επίση πολύ σημαντικέ προσπάθειες προκειμένου να διεκπαιρεωθούν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Όπως γνωρίζετε, το θέμα της, των εξαγωγικών φόρων και η αντιμετώπιση του αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι θα υπερκεράσουμε το συντομότερο δυνατό τις, ε, τους ενδιασμούς των συμβαλωμένων μερών για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΑΝ, ε, χρησιμοποίησαμε τη διμερή προσέγγιση και μάλιστα είχαμε δύο ε, γύρους διαπραγματεύσεων για την ε, σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Σιγκαπούρ και έπονται συμφωνίες με το Βιετνάμ και κατά πάσα πιθανότητα με την ε, Μαλαισία. Φυσικά, ο πότερος στόχος μας είναι μια περιφερειακή συμφωνία. Η Συμφωνία ελεύθερη Εμπορίου με την Κορέα μας χρησιμεύσε ώστε να μάθουμε, να πειραματιστούμε και να αντιληφθούμε καλύτερα τις συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας, κρατώντας ε, πολύ επικοδομητικό, στενό και συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διμερή ρήτρα διασφάλισης. Τον Απρίλιο, μάλιστα, στείλαμε στο Συμβούλιο προτάσεις για την υπογραφή προσωρινή εφαρμογή και την σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Μάλιστα προλιάναμε το έδαφος ώστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να αναλύσει το θέμα αυτό πριν την αναμενόμενη προσωρινή του εφαρμογή στα τέλη του έτους. Στο χώρο της Ασίας και πάλι Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εξαμήνου έγιναν δύο γύροι διαπραγματεύσεων τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ινδία. Συμφωνία με τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω όλε οι συμφωνίε με μεγάλε οικονομικέ συνέπειε, οι διαπραγματεύσει είναι περίπλοκε, παρόλο που υπάρχει δεδηλωμένη πολιτική βούληση και από τι δύο πλευρέ, γιατί είναι πεπισμένε ότι μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει ένα τεράστιο εμπορικό δυναμικό. Η ενίσχυση και η σύσφυξη των σχέσεων με την Κίνα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση στις αγορές, στις επενδύσεις και την πνευματική ιδιοκτησία αποτέλεσαν ε, προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Μάλιστα το Μάιο ε, έλαβε χώρα η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κίνας και έγινε μια απόπειρα επανισορρόπησης των διμερών σχέσεων. Επίσης θέλουμε να σημειωθεί απαραίτητη πρόοδος ώστε να μπορέσει και η Κίνα να προσχωρήσει στη Συμφωνία Δημοσίων ε, Προμηθειών του ΠΟΕ. Πριν από λίγε εβδομάδες έλαβε χώρα και διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Πακιστάν προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερο εμπορικό άνοιγμα τη χώρα, αυτή στα πλαίσια της μεταρρύθμιση του κανονισμού SPG. Σε ό,τι αφορά τι διμερείς μα ε, ε, σχέσει με τη Ρωσία που είναι στρατηγικό εταίρος μα. Καταρχήν, συμφωνούμε με την άμεση ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, καθώς και σε ένα ευρύ και αποτελεσματικό πλαίσιο νέων εμπορικών συμφωνιών στα πλαίσια μιας νέας συμφωνίας. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα για το εγγύς σε ό,τι αφορά τη χώρα αυτή. Από την άλλη πλευρά, ο νέος πρόεδρος Ουκρανίας ε, επανεπιβεβαίωσε την προσήλωσή του στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν ε, απτές ε, ε, την πρόοδο στα θέματα αυτά και στις ε, διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις ε, διατλαντικές σχέσεις, η, Ευρωπαϊκή, η Προεδρία της ε, Ισπανίας είναι υπέρ τη σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων με, την, με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Βέβαια, αναβλήθηκε η διάσκεψη κορυφή του Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, προχωρήσαμε στην μετατροπή του Διατλαντικού ε, Οικονομικού Συμβουλίου στο σε βασικό φόρουμ συνεργασίας και αριθμιστικής και στρατηγικής και μετά από συναντήσεις του Επιτρέπου Ντεγκούχτ με τον ε, ε, συμπρόεδρο Φρόμαν έγινε σημαντική πρόοδος στα πλαίσια αυτής της μετατροπής και μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να προσδιοριστεί το πρόγραμμα του ΤΕΚ μέσω και βράχη πρόθεσμα προκειμένου να τηρηθούν οι προτάσεις μας για στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και από τις δύο πλευρές. Έχουμε επίσης προχωρήσει σημαντικό όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια ευρύ οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Και στο δεύτερο εξάμενο αυτής της χρονιάς θα αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί βάσει των, της γραμμής που καθορίστηκε στην αρχή της εντολής. Με την Ιαπωνία επίσης έχουμε ενισχύσει τις προσπάθειές μας για τη σύσφυξη των εμπορικών μας σχέσεων μαζί της και θα ξεκινήσουμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας πριν καταλήξουμε σε αποφάσεις. Τέλος, για να τελειώσω με τις διμερείς σχέσεις, θα αναφερθώ στι συμφωνίες οικονομικής σύνδεσης με χώρες της Αφρικής, Καρυβικής και Ειρηνικού. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 6 από τις 8 τέτοιες συμφωνίες που σας ανέφερα πριν τον Μάγιο είχαμε το πρώτο μεικτό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Καριφόρουμος στα πλαίσια της διμερούς διάσκεψης και μάλιστα χτες και προχτές είχαμε το μεικτό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ. Η Ισπανική Προεδρία έκανε προσπάθειες να επικεντρωθεί στις ε, πρωτοβουλίες αυτές με τις χώρες ΑΚΕ προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη και η περιφερειακή ολοκλήρωση. Τώρα περνάμε σε θέματα οριζοντίου χαρακτήρα. Και εδώ θα αναφερθώ στη στρατηγική μα για την πρόσβαση στι αγορέ. Την 1η Ιουνίου που μα πέρασε, οργανώσαμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ισπανική Εργοδοσία και την Business Europe ένα πολύ ενδιαφέρον που στέφθηκε με επιτυχία μάλιστα σεμινάριο στη Μαδρίτη, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στην ενισχυμένη μα στρατηγική. Θεωρούμε ότι η μελλοντική εμπορική πολιτική μα πρέπει να δώσει ρόλο κλειδί στην ε, στρατηγική μα όσον αφορά την πρόσβαση στι αγορέ ή στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια, τις δημόσιες προμήθειες ή τα δικαιώματα πνευματική ε, ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά τους στόχους μας για τη στρατηγική του 2020. Όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων για την πνευματική ιδιοκτησία, έχουμε προχωρήσει πολύ αυτό το εξάμεινο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μας για την ε, συμφωνία την εμπορική κατά της ε, παραποίησης. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε τρεις γύρους διαπραγματεύσεων και ο τελευταίος γύρος θα λάβει χώρα το, στην Ελβετία την επόμενη εβδομάδα. Και ελπίζουμε ότι με τις διαπραγματεύσεις αυτές τις οποίες ενεργά συμμετείχε η Ισπανική Προεδρία στους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στην κοινή εμπορική πολιτική θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Επίσης, για να βελτιωθεί η πρόσβασή μας σε εξωτερικές αγορές, η Ισπανική Προεδρία έχει προωθήσει την εκπόνηση ενός εγχειριδίου στήριξης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται από τις διαδικασίες εμπορικού προστατευτισμού από τρίτες χώρες. Ήδη υπάρχει το εγχειρίδιο αυτό και θα επιτρέψει στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να αντιδράσουν με ελαστικότητα και ευελιξία στι περισσότερε ε, περιπτώσει και να γνωρίσουν καλύτερα τι βοήθεια μπορούν να έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τώρα και δύο σημαντικοί βιομηχανικοί τομείς Ευρωπαϊκή Ένωση που εξετάστηκαν ειδικά από την Επιτροπή εμπορική πολιτική, φαντουργία, Χαλιβουργία και άλλων βιομηχανικών προϊόντων που ονομάζουμε Επιτροπή STIS από τα αρχικά στα αγγλικά. Πρόκειται για τους ε, τομείς της κεραμικής και της επικοινωνίας για τις οποίες έχουμε ε, δύο ε, συγκεκριμένα στοιχεία όπου περιλαμβάνουμε όλες τις ευκαιρίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που τίθεται όσον αφορά την επέκταση των αγορών μας σε τρίτες αγορές. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω την προτεραιότητα που δώσαμε το εξάμεινο της Προεδρίας μας στην ενίσχυση για το εμπόριο. Εδώ πέρα πρόκειται για την οικονομική ανάπτυξη και για τη μείωση της ένδυας στις υπονάπτυξη χώρες. Δώσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνική αρρωγή σχετικά με το εμπόριο και τώρα θέλουμε να ασχοληθούμε με την βελτίωση της ποιότητας της αρρωγής μας αυτής. Πολύ σύντομα, ε, επευκαιρία της συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών για την αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το σημαντικό ρόλο που παίζει η αρρωγή αυτή στο εμπόριο. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας επίσης εκπονήσαμε και οθετήσαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα χρησιμοποιηθούν στη συνάντηση αυτή που θα λάβει η χώρα το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Όσον αφορά πάντα το εμπόριο, όπως λένε και οι στόχοι του προγράμματός μας, ε, προωθήσαμε και διαπραγματεύσεις όσον αφορά την Διεθνή Συμφωνία για την Εμπορία Όπλων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ετοιμάσαμε μία συγκεκριμένη δομή με ένα πρόχειρο για να πετύχουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μας όσον αφορά ε, τη συμφωνία που περιμένουμε για το 2012. Για τις διαπραγματεύσεις τώρα που έγιναν στην ομάδα εξαγωγών και πιστώσεων του ΟΣΑ, οι ομάδες που συμμετέχουν μετά μάλιστα από την οικονομική κρίση από την επλήγη το Προεδρείο, η Ισπανική Προεδρία έπαιξε επίσης ένα πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο. Ένα κατακλείδι. Λίγο πολύ αυτά είναι τα αποτελέσματα του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας στον εμπορικό τομέα. Ένα εξάμεινο που αναμφίβολα ήταν περίπλοκο και δύσκολο εξαιτία των θεσμικών και οικονομικών ε, εξελίσεων που είχαμε. Αλλά μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι για μας ήταν τιμή που ασκήσαμε την ε, Προεδρία κατά το εξάμεινο αυτό. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του στην τεράστια αυτή πρόκληση που αντιμετωπίσαμε. Βέβαια, οι υποχρεώσει μα δεν σταματάνε εδώ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στα πλαίσια του, των τριών προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου οι εμπορικές συναλλαγές μας να ε, μπορούν να προχωρήσουν και να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας και της απασχόλησης μέσα σε ένα ε, πολυμερές πλαίσιο με σαφείς κανόνες. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο στόχο μας αυτό, μια που αποτελεί όργανο κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διεξοδικότατη παρουσίασή σας για τα όσα έπραξε η Ισπανική Προεδρία για, την, για, το, για τη διεθνή εμπορική πολιτική και για τα όσα κάνατε και εσείς αυτό το εξάμεινο. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη. Ο Παύλο έχει καταρχήν το λόγο από το ΕΛΚ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Ισπανίδα Υφυπουργό, την κυρία Ράνσα και χαίρομαι ιδιαίτερω πολλών δεμάνων που είμαστε και συμπατριώτες. Ο πρόεδρο τη Ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε ω ικανοποιητική την Ισπανική Προεδρία. Θα προτιμούσε να την αποκαλούσε επιτυχημένη, αλλά μια και ήταν αρκετά πολυτάραχη αυτή η μήνε, σίγουρα αποσπάστηκε η προσοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση από του αρχικού στόχου τη Ισπανική Προεδρία και εντοπίστηκε αλλού. Νομίζω ότι ω προ πολλού στόχου τη ε, Ισπανικής Προεδρίας, το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιτυχημένο. Ξεπεράσετε το μέσο όρο σε πάρα πολλού τομεί. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την σύναψη εμπορική συμφωνία με το Περού και την Κολομβία, που προβλέπουν απελευθέρωση των συναλλαγών σε τομεί βιομηχανικών προϊόντων, αλληλεία γεωργικών προϊόντων, υπηρεσιών, επενδύσεων και ε, ξεκινά πολιτικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα κέριο σημείο της συμφωνίας αυτής. Επίσης, ε, ολοκληρώθηκε μια συμφωνία σύνδεσης με, μια με την ε, Κεντρική Αμερική. Πολύ σημαντική συμφωνία αυτή που ανοίγει ένα το φάσμα ευκαιριών και για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και για την κεντροαμερικανική οικονομία. Επίσης, ανοίγουν οι προοπτικέ για τη σύναψη συμφωνία ε, σύνδεση και με το Μερκοσούρ. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να προωθήσουν αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία. Έχουμε και το μηχανισμό επενδύσεων στην ε, Λατινική Αμερική. Εντυπωσιακή ήταν η πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία και με τον Καναδά. Πολύ ε, εντυπωσιακή αυτή η πρόοδο και θα είναι πολύ φιλόδοξη συμφωνία και αποφελή και για τι δύο πλευρέ. Επίση, προχώρησαν οι διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε με την Ινδία και τη Σιγκαπούρη. Σε ό,τι αφορά την διμερή ρήτρα διασφάλιση ε, τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κορέα, σα ευχαριστώ για την ειδική μνήμα που κάνατε Τη έκθεση μου. Θα ήθελα όμω να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά και θερμότατα την Ισπανική Προεδρία για τη βοήθειά τη. Βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα, υπήρχαν και κάποια σκοτεινά σημεία. Δεν υπήρξε πρόοδο, για παράδειγμα, στι διαπραγματεύσει ε, τη εμπορική τη Ντόχα. Πρόοδο αναμένεται μόνο μετά τα τέλη του 2011. Επίση, δεν είχαμε κανένα νέο μέλο στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Ούτε είχαμε κάποια πρόοδο στι νέε συμφωνίε ε, οικονομική σύνδεση και ήταν πολύ άτολμες οι πρωτοβουλίες σε σχέση με αυτά που μας είχε εξαγγείλει στις 27 Ιανουαρίου ο Υπουργό Σεμπαστιάν. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση του προστατευτισμού, προκειμένου να επιτύχουμε όλο και ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Εκεί δυστυχώς υστερήσαμε σε σχέση με τους στόχους. Ούτε ήταν πολύ φιλόδοξες ε, οι προσπάθειες που έγιναν σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Περιμέναμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και περισσότερα επιτεύγματα στους τομείς αυτούς από την Ισπανική Προεδρία. Δυστυχώς αποτερματώθηκε από ό,τι φαίνεται και η διαδικασία της Βαρκελόνης. Χρειάζεται λοιπόν να επιτείνουμε τις προσπάθειες μας εκεί. Όπως σας είπα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ε, χαρακτήρισε ε, ικανοποιητική την Ισπανική Προεδρία. Για τις εμπορικές όμως ειδικά σχέσεις, η Ισπανική Προεδρία ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, ήταν πολύ επιτυχημένη και θα ήθελα να σας συγχαρώ γι' αυτό. Ο κύριος Μενέντες, Δελβάγε. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Υφυπουργέ, κύριε Μπονέτ. Ίσως ε, θα φαινόταν άπρεπο από πολιτική άποψη ένας Ισπανός και μάλιστα από το κυβερνόν σώμα να σας ε, απευθύνει θερμούς χαιρετισμού ε, και ευχαριστίες ε, πιο έντονες από ό,τι ο κύριος Σάλβα. Εντάξει, μπορεί να είναι ε, πολιτικός άπρεπο, αλλά παρόλα αυτά θα επιτρέψω στον εαυτό μου αυτή την, αυτή την παρατυπία. Όπως είπε και ο κύριος Σάλβα που επίσης ήταν εγκομιαστικός απέναντι στην Ισπανική Προεδρία και εγώ είμαι ενθουσιασμένος από τα επιτεύγματα της Ισπανικής Προεδρίας και θα ήθελα να σας, συγχαρώ θερμά. Θα ήθελα να πω στον Παύλο Σάλβα και φαντάζομαι συμφωνεί μαζί μου ότι το, το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις Ντόχα δεν έχει σχέση με τις προσπάθειες ούτε της Ισπανικής Προεδρίας ούτε με τη δράση του Πρόεδρου Βαν Ρομπόη. Είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις Ντόχα και θα χρειαστεί πολύ χρόνος για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις τώρα και αν υπάρξει δυνατότητα και δεύτερο γύρο θα συνεχίσω αργότερα. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά, αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με, το Μερκοσούρ. Θα γνωρίζετε κύριε Υφυπουργέ ότι ένα τμήμα της Επιτροπής μας θεωρεί ότι εξαιτία των αλλαγών της παγκόσμιας οικονομίας η διαπραγματευτική εντολή του Δεκεμβρίου του 2009 ίσως ε, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί γιατί είναι κάπως παροχημένη. Γνωρίζετε και το επισημάναμε και στον Επίτροπο Ντεγκούχτ ότι η θέση της Επιτροπής ε, είναι αντίθετη, δηλαδή θεωρεί ότι η διαπραγματευτική εντολή περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγκυα, ε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες ε, που διαμορφώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία εξαιτία της κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω μια ερώτηση. Εσείς τι γνώμη έχετε, γιατί Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο διαφωνούν ως προς αυτό. Συμφωνείτε να γίνονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων για απολογισμό της κατάστασης. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε μια αισιοδοξία ως προς την ε, επαναφορά του Εκουαντόρ στην ε, διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Σύνδεσης, όπως έγινε και με την Κολομβία και το Περού. Εγώ έχω και άλλε ειδήσει. Άκουσα ότι η Βολιβία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, θεωρεί τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγικής σημασίας. Μάλιστα, οι τελευταίες ε, ειδήσει ε, μα μεταφέρουν ότι πολύ πιθανό η χώρα αυτή, η Βολιβία, να ακολουθήσει το δρόμο του Εκοντόρ και πολύ σύντομα να συμπεριληφθεί στις χώρες της κοινότητας των Άνδεων που τάσσονται υπέρ αυτή τη συμφωνία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ούτε εκ μέρους βολιβία, Βολιβίας, ούτε εκ μέρους Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής ότι θα εγκαταλειφθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης που γίνεται με ολόκληρη την κοινότητα των άνδρων. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Παρόλο που τα ισπανικά είναι πολύ όμορφη γλώσσα, αλλά δεν είναι η μόνη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας ακούσουμε και κάποιον άλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, καλώ ήρθατε. Μετά τις παρατηρήσεις των Ισπανών συναδέλφων, εκδεξιών και ξεβονίμων, θα ήθελα και εγώ να αποφαθώ, παρόλο που δεν είμαι Ισπανός, αλλά κανένας δεν είναι τέλειος, όπως ξέρετε. Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τις επιτυχίες σας ε, στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας. Ομολογούμε ότι η Προεδρία αυτή έλαβε χώρα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέπεσε με την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας οπότε χρειάστηκε να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες και στις νέες διαδικασίες ενισχυμένης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε ιδιαίτερος από την πλούσια εμπειρία που είχαμε για πρώτη φορά με την Ισπανική Προεδρία με τη συνθήκη της Λισαβόνας διαπιστώσαμε ότι σημειώθηκε πρόοδο στι διαπραγματεύσει με τις χώρες της Λατινική Αμερικής, το Μερκοσούρ, την Καραϊβική και πραγματικά σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε εσά αυτά τα επιτεύγματα, παρόλο που εκκρεμούν ακόμη κάποια προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε ένα άλλο θέμα, μερικά από αυτά αναφέρθηκαν ήδη από τον συνάδελφο Σάλμπα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στι εμπορικέ διαπραγματεύσει του γύρου τη Ντόχα. Χθε είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τον επίτροπο Κάρελ Τεγκούχτ και ήταν αρκετά αισιόδοξο. Βέβαια, εξέφρασε την επιθυμία του να επιδείξουν και οι Αμερικανοί μεγαλύτερο πνεύμα πρωτοβουλία για να προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την αισιοδοξία του αρμόδιου επιτρόπου. Πιστεύετε ότι του χρόνου θα τελεσφορήσουν και θα δεκπεραιωθούν οι διαπραγματεύσει τη Ντόχα. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την παράταση του ισχύοντος κανονισμού SPG-SIN. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε παράταση χωρίς ουσιαστική όμως αναθεώρηση του κανονισμού. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο καλούνται να το εγκρίνουν. Από ό,τι ξέρω όμως κάποιες χώρες είναι υπέρ ε, μιας αλλαγής και αναθεώρησης αυτού του κανονισμού. Εσείς τι γνώμη έχετε. Και Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι έγινε μια παρουσίαση της στρατηγικής για την κοινή εμπορική πολιτική ενόψη της στρατηγικής του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, από την εμπειρία που αποκομίσατε το τελευταίο εξάμεινο, θα μπορούσατε να μου αναφέρετε τις πέντε προτεραιότητες που είναι κατά τη γνώμη σας σημαντικές και καλό θα ήταν να επιδιωχθούν από τις επόμενες προεδρίες προκειμένου να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ. Εγώ δυστυχώς δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας για πολλά και διάφορα θέματα. Και έχω πολλές ανησυχίες για το θέμα της επανάληψης ε, των διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ και για τις συμφωνίες με το Περού και την Κολομβία. Γνωρίζετε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ύφεση, με απώλεια θέσεων απασχόλησης, με αύξηση της ανεργίας, αποσταθεροποίηση του, του λαού. Το ξέρετε και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες η κατάσταση είναι δεινή. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς επιλέξαμε για να διαπραγματευτούμε πλεονεκτήματα ε, για τις χώρες Λατινικής Αμερικής και αυτό με ανησυχεί. Οι συμφωνίες Περού και Κολομβίας θα αποσταθεροποιήσουν ένα τμήμα των ε, υπερπόντιων διαμερισμάτων της Γαλλίας και αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη γιατί θα διεκδικήσουμε κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που θα έχουν τα διαμερίσματα εξαιτία των εμπορικών συμφωνιών με το Περού και την Κολομβία. Επίση. Ε, υπάρχει τεράστιο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε δίνη κατάσταση. Γιατί με τις συμφωνίες αυτές η, αυξήσεις, ε, η αύξηση των εισαγωγών του βοήου κρέατος φτάσει στο 65% και 25% του κρέατος πουλερικών. Παρόλο που οι χώρες αυτές δεν τηρούν ούτε τις κοινωνικές ούτε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που επιβάλλουμε στην εγχώρια μας ε, γεωργία και κτηνοτροφία. Εγώ δεν είμαι υπέρ άκρα του προστατευτισμού, αλλά θα πρέπει να είμαστε ευφύς και δίκαιοι. Δεν θα πρέπει στην ε, ευρωπαϊκή μας πολιτική να είμαστε προσιλωμένοι σε ένα θέμα και να διαφορούμε για τα κοινωνικά περιβαλλοντικά θέματα αλλού ή τι αντίκτυπο έχουν σε ό,τι αφορά την απώλεια θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη τέτοιου είδου εμπορικέ συμφωνίε. Και τέλο, σε ό,τι αφορά την Ένωση για τη Μεσόγειο, προ το παρόν είναι αποτυχία αυτό το εγχείρημα. Βέβαια δεν φταίει μόνο η Ισπανική Προεδρία γι' αυτό, φταίει και η κρίση στην ε, Μέση Ανατολή. Δημιουργήθηκαν πολλές προσδοκίες με την Ένωση για τη Μεσόγειο, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε δύο τομεί. Καταρχήν στον πολιτικό, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα της ε, επίλυσης ε, του Μεσανατολικού, να ταχθεί πιο ενεργά υπέρ της ε, ειρήνευσης εκεί και να αναλάβει κινδύνους και για το οικονομικό θέμα που επίσης είναι σημαντικό. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία για τα όσα έκανε παρά την ε, σοβαρότητα της κρίσης που περνούμε. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει πολλές επιτυχίες και ακόμη υπάρχει ε, χρόνο στις λίγες τελευταίες μέρες που απομένουν στην ε, Ισπανική Προεδρία να στείλει ένα ισχυρό, ηχηρό μήνυμα προς την επόμενη Προεδρία. Πιστεύω ότι εμείς που εμπλεκόμεθα στον τομέα του εμπορίου έχουμε καθήκον να ζητήσουμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από το Συμβούλιο στις μεγάλες ε, αποτυχίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, την έλλειψη οικονομικής πολιτικής. Δεν μπορεί να θέλεις εμπόριο, δεν μπορεί να θέλεις κοινωνικές δραστηριότητε. δεν μπορεί να κάνεις τίποτα που να ενισχύει την ε, ανάπτυξη στη χώρα σου εάν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, οικονομική πολιτική και δεν μιλώ μόνο για νομισματική πολιτική. Τώρα επιτέλους ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Αν λοιπόν ε, αυτό το αίτημα καταστεί πιο σαφές λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις, α, τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι θα ήταν καλό. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εναρμόνισης των τελωνιακών δασμών. Όπως είπε και ο Επίτροπος Δεκούχτ εχθές, υπάρχει κάποια εναρμόνιση, αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν ξέρει πολύ καλά ότι η εναρμόνιση ισχύει σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά όχι σε επίπεδο ελέγχων, σε επίπεδο επιθεωρήσεων, Υπάρχουν ε, κάποια τελωνιακά, κάποιε τελωνιακέ υπηρεσίε που λειτουργούν σωστά και, και εμποδίζουν την εισαγωγή κύβδηλων προϊόντων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και κάποιε υπηρεσίε που δεν λειτουργούν σωστά. Λοιπόν, ε, του ελέγχου, πρέπει να τους εντείνουμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένη από την δουλειά που έκανε η Ισπανική Προεδρία σε ό,τι αφορά και την συμφωνία για την παραχάραξη και για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ελπίζω ότι αυτή η υποστήριξη και η ελπίδα να είναι ένα ηχηρό μήνυμα και για το μέλλον. Και ένα τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε. Ε, ήδη αναφερθήκαμε και σε παλαιότερε συνεδριάσει στο θέμα αυτό. Η Ευρώπη πάει πολύ γρήγορα προς πολλές ε, συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Εντάξει, όταν έχουμε να κάνουμε με μικρέ χώρε, ωραία, καλώ ε, υπογράφονται αυτέ οι, οι συμφωνίε για να βοηθήσουμε τις, ε, και τι δικέ μα τι εταιρείε και τι εταιρείε τη άλλε χώρε, έτσι σε μια βάση αμοιβαιότητα. Αλλά όταν μιλούμε για χώρες όπως η Ινδία ή άλλες που αναφέρθηκαν, ε, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πρόωρο. Οπότε και πάλι, μια που είναι και φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της προεδρίας σας, θα ήθελα να σας ζητήσω και από σας και από το Συμβούλιο να δώσετε περισσότερη προσοχή στον κανονισμό για τον καθορισμό της προέλευσης για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει μειονέκτημα έναντι άλλων χωρών, όπως η ΕΠΑ, ας πούμε, εφόσον υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε, ο Τζον Χίγγινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η Ισπανική Προεδρία προέδρευσε μιας περίοδου 6 μηνών όπου είδαμε το μεγαλύτερο δυνατό ε, κερδοσκοπικό παιχνίδι από κερδοσκόπους, από hedge funds έναντι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ήταν το χειρότερο παράδειγμα. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία επίσης πλήγησαν από αυτούς. Εσείς τώρα ως υπουργό Εμπορίου θα πρέπει να ξέρετε ότι όσο περισσότεροι πόροι απορροφώνται από αυτά τα παράσιτα των οικονομικών αγορών, τόσο πιο βαθιά θα είναι η οικονομική κρίση στον τομέα των κατασκευών και της υπηρεσίας μόνο και, μόνο, και των υπηρεσιών, επειδή μόνο και μόνο επειδή τόσα, τόσοι πολλοί δημόσιοι πόροι που θα έπρεπε να, ε, να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες πάνε για να, να ξεπληρωθούν ε, οι κερδοσκόποι των αγορών. Να σας ρωτήσω λοιπόν, εσείς πώς δικαιολογείτε, πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι η Ισπανική κυβέρνηση, όπως και η δική μου κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, έχει κεφαλαιοποιήσει ε, έναντι των ε, ε, κερδοσκόπων. Τώρα επιτίθεστε ε, με ισχυρότατο τρόπο στις συντάξεις, στο επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων και πώς δεν έχετε ακόμη ε, αλλάξει το σύστημα. Πώς δεν έχετε βάλει τους, τους κερδοσκόπους ε, στη θέση τους. Γιατί πραγματικά οι συνέπειε είναι καταστροφικές και για το εμπόριο και για την οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερο, να σας ρωτήσω και πάλι. Σε σχέση με την ε, συμφωνία για ελεύθερο συνεργό με την Κολομβία και το Περού, πώς δικαιολογείτε το ότι αντιτίθεστε σε όλα όσα έχουν ζητήσει οι, τα συνδικάτα στην Κολομβία, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν το ανθρώπινα δικαιώματα, το, τους, ε, ε, τους γηγενείς ε, που δεν ήθελαν αυτή την, αυτή την συμφωνία. Συνάπτω συμφωνία με μια τέτοια χώρα που παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών της κατά τη διάρκεια της δικής σας ε, προεδρίας ανακαλύφθηκαν αυτοί οι τάφοι μαζικών ενταφιασμών. Πώς μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε ως οτιδήποτε άλλο πέρα από το ότι απλώς ε, βοηθάτε ε, την κυβέρνηση της Κολομβίας που κατηγορείται για όλα αυτά τα εγκλήματα ή μήπω το ενδιαφέρον, τα συμφέροντα των ε, ισπανικών επιχειρήσεων μπήκανε μπροστά από τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπερτέρησαν. Ε, επίσης, σε σχέση με τους, ε, τις συμφωνίες με τις χώρες της Κεντρικής, Αμερική, με τις, της Κεντρικής Αμερικής, πώς ακριβώς δικαιολογείται την συμφωνία με, με την Ονδούρα, μια πολύ στημένη διαδικασία που ξεκίνησε και με πραξικόπημα. Τι σήμα δίνουμε σε σχέση με αυτά που είναι διατεθειμένη να κάνει η Ευρώπη για να εξασφαλίσει τέτοιου είδους συμφωνίες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τις απαντήσεις και τα σχόλια της Υφυπουργού. Εκ μέρου τη Ισπανική Προεδρία, λοιπόν, κυρία Ιράντσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις από το ΕΛΚ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και για τη στήριξή σας στην Ισπανική Προεδρία. Εκεί οφείλεται και η επιτυχία της Ισπανικής Προεδρίας. Συγχρόνως βέβαια να γνωρίζουμε, όπως είπε και ο κ. Σάλμπα πολύ σωστά, ότι υπάρχουν κάποια θέματα όπου όσο και αν προσπαθήσαμε δεν ήταν δυνατόν να πετύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα γιατί απλά δεν ήταν στο χέρι μας να τα πετύχουμε. Πολύ θα θέλαμε να είχαμε δει πρόδους και στο γύρο της Ντόχα, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κύριος Άλμπα, υπάρχουν εδώ προϋποθέσεις πολύ σημαντικές, και έτσι απαντάω και σε άλλες ερωτήσεις που μου υποβάλατε, ότι υπάρχουν θέσεις πολύ μεγάλων και σημαντικών χωρών, τόσο αναπτυγμένων όσο και αναδιόμενων, που δεν βοήθησαν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ήταν αδιάλακτα σε μερικά ζητήματα. Όσο δεν προχωράει λοιπόν ο γύρο τη Δόχα, δεν θα ξέρουμε ποια θα είναι και η τελική θέση των ΗΠΑ. Είμαστε όμω αισιόδοξοι, γιατί η επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει τον 20 στο Τορόντο μπορεί να μα δείξει κάποια πρόοδο. Έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις του κυρίου Μενέντεθ. Τι γνώμη έχουμε για την εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ. Εμείς πιστεύουμε ότι η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή πριν από μερικά χρόνια για να προχωρήσει σε με την Μερκοσούρ εξακολουθεί να ισχύει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγέ, αλλά όπως είπε και κάποιο άλλο εδώ, πραγματικά αυτά τα οποία μα απασχολούσαν πριν από μερικά χρόνια εξακολουθούν να μα απασχολούν και να μα ανησυχούν. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο νέο στάδιο που βρισκόμαστε και έτσι σε αυτήν τη συνάντηση θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση. Ανάλογα θα δούμε αν πρέπει να αλλάξει εντολή ή όχι. Πάντως αν δεν γίνει αυτός ο πρώτος γύρος δεν θα το ξέρουμε. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι θα ήταν καλό να μπορέσουμε να ενημερώσουμε λιγάκι τις μελέτες που γίνουν για τον αντίκτυπο επιπτώσεων. Όσον αφορά τώρα τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Ευτυχώς ξαναρχίζουν διαπραγματεύσεις, Ξανάρθαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Ισημερινός και η Βολιβία. Για τη Βολιβία νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε προσωπική εκτίμηση, γιατί η Βολιβία έχει κάθε συμφέρον να επανέλθει στο, στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων γιατί οι συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού που ολοκληρώθηκαν δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε και τον Ισημερινό και τη Βολιβία για να αρχίσουν να ισχύουν οι συμφωνίες αυτές που είναι σημαντικές για αυτές τις χώρες καταρχήν. Έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις του κύριου Καζάκ για το θέμα του γύρου της Ντόχα. Βέβαια, πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε βήματα προς τα μπρος θα πρέπει να βασιστούν στις πρόοδους που πετύχαμε το 2008. Πάντως στον Καναδά μας δίνεται μια καλή ευκαιρία για να δούμε τις θέσεις των διαφόρων μεγάλων χωρών σε αυτό το τομέα. Έρχομαι τώρα στον τομέα του SPG. SPG. Ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία προκειμένου να τροποποιηθεί ο κανονισμός αυτός. Εμείς πιστεύουμε για να είναι πιο δίκαιο το σύστημα για τις χώρες οι οποίες εποφελούνται από τις γενικευμένες προτιμήσεις θα έπρεπε να αναθεωρηθούν τα οικονομικά κριτήρια και να επιλέξουμε καλύτερα τις χώρες που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη συμφωνία. Για να μην αποκλείουμε αναδιόμενες χώρες. Επίσης, πρέπει να δούμε αν θα συμπεριλάβουμε και ειδικά προϊόντα. Επίσης, να αναθεωρήσουμε και το κριτήριο ε, του ευάλωτου μιας χώρας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα κριτήρια και για το σύστημα SPG και για το SPG-SYN, συμπεριλαμβάνοντας τη ρήτρα της χώρας καταγωγής. Όσον αφορά τις προτερότητές μας στο καθορισμό της στρατηγικής 2020 στον εμπορικό τομέα, Βάσει του εγγράφου της 3ης Μαρτίου της Κομισιόν και του εγγράφου που βασίζεται στη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Ιούνιο και που θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουλίου. Βάσει λοιπόν των συμπερασμάτων αυτών θα συμπεριλάβουμε διάφορες προτεραιότητες. Ζητήσατε πέντε δεν ξέρω αν θα είναι πέντε ή τέσσερις, πάντως οι κυριότερες θα είναι πρώτον η ολοκλήρωση των πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται, κυρίως εκείνες που έχουν μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις στον πόριο. Δεύτερον, θα έλεγα καλύτερη βελτίωση των συμφωνιών που ήδη υπάρχουν, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στους μη δασμολογικούς φραγμούς. Είναι πολύ σημαντικό. Σε όλο τον κόσμο μειώνονται οι δασμοί. Τρίτον, μεγαλύτερη προσοχή σε πρωτοβουλίες εμπορικού ανοίγματο σε διάφορους τομείς που έχουν μέλλον, όπως είναι η πράσινη τεχνολογία, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και οι προτάσεις για τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομούς με μεγάλο δυναμικό. Επίσης, ως προτεραιότητα, εμείς βάζουμε και τον διάλογο υψηλού επίπεδου μετέρους κλειδί για θέματα όπως είναι η πρόσβαση στις αγορές, ρυθμιστικό πλαίσιο, ισορροπίες και ανισορροπίες, ενέργεια, κλιματικές αλλαγές, πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ένδια, εκπαίδευση και ανάπτυξη. Και βέβαια, ενίσχυση του διαλόγου με τις Ηνωμένε Πολιτείες, διάλογος υψηλού επίπεδου με την Κίνα και ενίσχυση των σχέσεών μας με χώρες όπως είναι η Ιαπωνία και η Ρωσία. Φυσικά υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στις αγορές. Θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες, προκειμένου να πετύχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, στις ξένες αγορές. respondiendo a las cuestiones eh, απατώντας ε, στις ερωτήσεις της κυρίας Αρνές για το Μερκοσούρ. Θεωρούμε τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, που σίγουρα θα είναι χρονοβόρα και θα απαιτήσει πολύ σκληρές προσπάθειες, με βάση τη διαπραγματευτική εντολή που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφωνία με το Μερκοσούρ θα εξασφαλίσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, πλεονεκτήματα, πολύ απτά ωφέλη από την συμφωνία αυτή. Για παράδειγμα, θα εξασφαλίσουμε πρόσβαση της ε, ευρωπαϊκής επιχειρή... Ε, ε, βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ήταν κλειστές οι αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά ευκαιρίες θα υπάρξουν και για τη χημική βιομηχανία, τη φαρμακευτική, τα καλλιτικά προϊόντα, την κλωστοϊφαντουργία και τη βιομηχανία υπόδησης. Θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά για πολλοί άλλους σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως είναι έλεα, ε, ειδήποτα, ίνι κτλ. Ε, ε έγινε και με τις... Ε, δείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Βέβαια, όλες αυτές οι συμφωνίες της νέας γενιάς είναι ευρύτατες και θα βρούμε και νέες ευκαιρίες και για επενδύσεις. Θα αποκτήσουμε κάποια βελτίωση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την προστασία των επενδύσεων. Θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανική παραγωγή και στις επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ωφέλη τεράστιες ευκαιρίες θα δημιουργηθούν και με τη Βραζιλία, σε, στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αγροπιστιστική βιομηχανία, γεωργία, κατασκευή, μηχανολογικά προϊόντα, μεταφορές. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι οι δημόσιες συμβάσεις, οι δημόσιες προμήθειες. Ε, το Μερκοσούρ μας έδειξε την προθυμία του να διαπραγματευτεί άνοιγμα σημαντικών τομέων δραστηριοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, θα έχουμε και τους Ολυμπιακούς ή το Μουντιάλ στη Βραζιλία, κάτι που θα ανοίξει τεράστιες ευκαιρίες για τις υποδομές. Υποδομές που μέχρι στιγμής ήταν κλειστές απέναντι στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και όλα αυτά θα γίνουν χάρη στην σύναψη αυτή τη συμφωνία. Πάντως είναι τεράστια πρόκληση που δημιουργεί αυτή η συμφωνία, αλλά και οι τεράστιε ευκαιρίε που θα διανοιχθούν για τι επιχειρήσει μα. Σε ό,τι αφορά την ευρωμεσογειακή διαδικασία, τη διαδικασία τη Βαρκελόνη και την Ένωση για τη Μεσόγειο, εκεί υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί παράγοντε που δυστυχώ εμποδίζουν την υλοποίηση πρόοδου στις οικονομικές πτυχές, στη σύναψη οικονομικών συμφωνιών με τις χώρες αυτές. Το πολιτικό υπόβαθρο είναι δυσχερές και παρεμποδίζει και το οικονομικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή, εκεί έχουμε σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δώσουμε όθηση στο εμπόριο του Νότου, στην ολοκλήρωση μεταξύ χωρών του Νότου, διαδικασία του Αγαδίρ. Υπάρχει μια δίλη πρόοδος εκεί. Επίσης θα πρέπει να αντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ε, για να ενισχύσουμε μια πολυμορφία των συναλλαγών και να προωθήσουμε μεγαλύτερη βιομηχανική και περιφερειακή ολοκλήρωση. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις της, του κυρίου Higgins από την ΚΟΕ, Α, συγγνώμη. Ξέχασα την κυρία Μουσκαρντίνη. Είναι πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας, κυρία Μουσκαρντίνη. Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και θα μας εμπνεύσουν ε, στην ε, μελλοντική μας εμπορική πολιτική, που είναι πολύ σημαντική για την ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας, κυρία Μουσκαρντίνη. Και επανέρχομαι στις ερωτήσεις του κυρίου Χίγκινς από την ΚΟΕ. Μας ρωτήσατε κύριε Χίγγινς γιατί συνθηκολογήσαμε μπροστά στους κερδοσκόπους και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκάλεσαν στο εμπόριο. Με βάση τα στοιχεία μας, το διεθνές εμπόριο, ξεκινώντας με το γενικό, αυξήθηκε κατά 25%. Το 25% είναι διόλου αμεληταίο ποσοστό πέρυσι μάλιστα, που ήταν η χειρότερη διαχειριστική χρήση από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για το Διεθνέ εμπόριο, μειώθηκε το ποσοστό σε 12, κατά 12%. Το εμπόριο όμως βοηθά την οικονομική ανάπτυξη, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και δίνει όθηση και στην απασχόληση. Και μάλιστα το εξωτερικό εμπόριο είναι αυτό που βοηθά περισσότερο να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να αναζωογονηθεί η οικονομία και η επαγγελματική δραστηριότητα. Το 2009 ο εξωτερικός κλάδος στην Ισπανία πρόσφερε 2,8 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης στο ΑΕΠ και το 2009 θα προσφέρει πάνω από 1,5% ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ. Η στρατηγική του 2020 είναι κάτι που θα συνεχιστεί και θα σφυριλατηθεί γύρω και από τον εμπορικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τα σχόλιά σας για τις συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού, σίγουρα όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ σημαντικά και ξέρω ότι συζητήθηκαν διεξοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα ε, και μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία μετέβη στην Κολομβία για να διαπιστώσει στην πράξη αν ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων. Βέβαια μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά ήταν ορατές ε, οι προσπάθειες που έγιναν και η που σημειώθηκε φαίνεται και από τις εκθέσεις της ΔΟΕ και από τις εκθέσεις του ΟΗΕ, αλλά και από τις μελέτες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στους τομείς που αναφέρατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα τη αηφόρου ανάπτυξη, όλα αυτά τα αναπτυξιακά ζητήματα αποτελούν ε, κεντρικό άξονα όλων των εμπορικών συμφωνιών νέα γενιά που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ομιλούμε καθόλου ούτε τα κοινωνικά ούτε τα εργασιακά δικαιώματα. Τη χάνουν ιδιαίτερη μεταχείριση στι νέε εμπορικέ μα συμφωνίε και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ την πρόοδο αυτή τη κατάσταση στο μέτρο που αρχίζει και εφαρμόζεται μια δεδομένη εμπορική συμφωνία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό για την εις και την ειλικρινέστατη απάντηση, αξιολόγηση για τα επιτεύγματα της Ισπανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχετε επιτυχία και σε αυτούς αλλά και σε άλλους τομείς στην ε, Ισπανική κυβέρνηση. Κλείνουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Επόμενη συνεδρίαση 13 και 14 Ιουλίου.